we painting in English? So, ladies and gentlemen, please be seated. Καθίστε παρακαλώ. Όσοι θέλουν να αποχωρήσουν, βεβαίω και μπορούν, αλλά γρήγορα παρακαλώ. So, να καλωσορίσουμε τον κύριο Γκούν Βερβάκε. Είναι Διεθνών Σύμβουλο ε, τη Υπηρεσία Εξωτερική Δράση για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την Αφρική. Θα μα ενημερώσει για τι πρόσφατε εξελίξει στην Αιθιοπία, το Σουδάν και το Νότιο Σουδάν. Θα θέλουμε, κύριε Βερβάκε, να μα ε, περιγράψετε τι πρόσφατε εξελίξει σε αυτέ τι χώρε. Ε, είδαμε το 2018 ο Άμπι Αμέντ ανέλαβε τα ενία της Αιθιοπίας. Ε, υπήρξαν σημαντικές μεταρρυθμίσεις ε, σε πολιτικό, οικονομικό, ε, και κοινωνικό επίπεδο, καθώ και στην εξωτερική πολιτική, όμω, ε, παραμένουν προκλήσεις όπως ε, κατέστη σαφές και από την, από την απόπειρα πραξικοπήματο την περασμένο μήνα. Θα ήθελα να μα μιλήσετε για την κατάσταση, τις επερχόμενε εκλογέ και για το πώ η Ευρωπαϊκή Ένωση συμβάλλει στο να στηρίξει την Αιθιοπία σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Το Σουντάν αποτέλεσε θέμα συζήτησης και στο Υπουργείο Εξωτερικών Υποθέσεων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 έχει τεθεί πλειονεφική στην κεφαλή του Ευρωπαϊκού Θεματολογίου εξαιτία της προσέγγισης ε, που ε, ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και θα ήθελα να τονίσω ότι στα τέλη της επόμενης χρονιάς η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, θα διοργανώσει την επόμενη διάσκεψη μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αφρικής εδώ στις Βρυξέλλες και θα είναι μια πολύ σημαντική στιγμή για να παγιώσουμε μια νέα, πιο πολιτική προσέγγιση κοινών συμφερόντων που ακολουθούμε από την περασμένη ε, τέτοια διάσκεψη στην Αβιτζάν. Και στο πνεύμα που πρότεινε ο κύριος Γιούνκερ με την ε, οικονομική διάσταση των σχεσιών μας αλλά και την πλευρά της ασφάλειας, κλιματικής αλλαγής, της μετανάστευσης και καθώς τώρα η Αφρική αποτελεί ε, κέριο παίκτη σε ό,τι αφορά τις ε, πολυμερείς ε, προσπάθειες και με τα χαρά θα επανέλθουμε στην Επιτροπή σας ε, όποτε μας το ζητήσετε. Μου, μιλήσατε να σας, μου ζητήσατε να σας παρουσιάσω την κατάσταση για την Αφρικανική Ήπειρο. Έχουμε αναπτύξει λοιπόν εξωτερική πολιτική ως προς την Αφρική με πολλούς ε, θεματικούς στόχους, ε, κλιματική αλλαγή, μετανάστευση, οικονομική πρόσβαση και σταθερότητα στο κέρας της Αφρικής. Όλα αυτά συνδέονται με αυτό. Και η Αιθιοπία αποτελεί πολύ σημαντική χώρα προς αυτό. Είναι μια πολύ σημαντική χώρα για, για εμάς ε, πάνω από 100 εκατομμύρια κατοίκοι, μια χώρα σε καθεστώς μετάβασης. Ξέρετε, ο Ταχάλε ανέλαβε και παρετήθηκε μετά το 2018 και μετά ανέλαβε ο Αμπί Αχμέτ. Είναι η πρώτη φορά που εξελέγει ένας ε, πρωθυπουργό που δεν προέρχεται από την εθνοτική ε, κοινότητα Τίγρεϊ και αυτό δείχνει μια τεράστια μεταστροφή της πολιτικής σκηνής ε, στην Αιθιοπία προέβη, όπως είπατε Πρόεδρε, σε σημαντικές ε, μεταρρυθμίσεις, επιστροφή των ε, αρχηγών της αντιπολίτευσης, απελευθέρωση πολιτικών κρατουμένων, ε, άνοιγμα των μέσων ενημέρωσης, υπήρξαν κάποιες προσεγγιστικές ενέργειες με την Ερυθρέα, τη γείτονα χώρα και σημαντικές οικονομικές μεταρρυθμίσεις επίσης. Αυτό βέβαια ανέδειξε δυνάμεις που είναι δύσκολο να τις ελέγξει κανείς. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να επιθέσουμε την προσοχή μας σε όλα αυτά τα ζητήματα. Ε, στρεφόμαστε προς μία ε, πιο ομοσπονδιακή προσέγγιση, αλλά υπάρχουν και εθνοτικές εντάσεις ε, μεταξύ των ευμέρους κοινοτήτων. Ε, προσφάτως, αυτές οι εντάσεις και μια πιθανή ε, πρόκληση αποτυπώθηκε στην δολοφονία ε, σημαντικών προσωπικότητων, ε, του επιτελάρχη ας πούμε του περιφερειακού, περιφερειακών στρατιωτικών δυνάμεων και του ηγέτη της περιοχής Αμάρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει πλήρως την, την ηγεσία και ο Επίτροπο Μίμητσα επισκέφθηκε την Μπέμπα και η υπατεκπρόσωπος Μογκερίνη καθώς και η ηγεσία της Επιτροπής και παρέχουμε όποια στήριξη μπορούμε προκειμένου αυτές οι μεταρρυθμίσεις ε, να μπορέσουν να υλοποιηθούν και από οικονομικής και από πολιτικής άποψης. 1,6 δις ευρώ έχουν ε, διοχετευτεί προς την Αιθιοπία για την αναπτυξιακή συνεργασία και μετά την επίσκεψη του Επιτρόπου Μίμητσα 100 εκατομμύρια επιπλέον χρηματοδότηση και στήριξη ε, αποφασίστηκε να διοχετευθούν για περαιτέρω στήριξη. Και από πολιτική άποψη ε, είμαστε διατεθειμένοι να τους ε, στηρίξουμε για τις εκλογές σε συνεργασία βέβαια με τις τοπικές αρχές. Η ανθρωπιστική κατάσταση εξαιτία όλων αυτών των εντάσεων είναι δύσκολη πάνω από ένα εκατομμύριο εκτοπισμένοι. Αποτελεί αυτό πραγματική πρόκληση για τις ε, οργανώσεις ανθρωπιστικής βοήθειας. Πρέπει να βρούμε την σωστή ισορροπία, γιατί όπως είπα υπάρχουν εντάσεις και πιέσεις. Και αυτό επηρεάζει και την ε, διαχείριση αυτού του προβλήματος ε, των ιστορικά εκτοπισμένων. Για το Σουδάν τη Δευτέρα. τη της ε, συνεδρίασης φίλη του Σουδάν ε, ακριβώς πριν από το ε, Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων και την επίσκεψη εκπροσώπου της Φιλανδίας εξ ονόματος της ΥΠΑ της εκπροσώπου είναι μια μοναδική ευκαιρία τώρα να ξαναμπεί σε, στη σωστή τροχιά ε, η χώρα μετά από 30 χρόνια της δικτατορίας Μπασίρ, ο οποίος ε, ανατράπει τον Απρίλιο με στρατιωτικό πραξικόπημα, όπως ξέρετε. Όμως ε, το πραγματικό σημείο πίεσης ήταν οι ειρηνικές διαμαρτυρίες που ξέσπασαν στη χώρα. Έχουμε λοιπόν μια πολύ καλή ευκαιρία. Πολιτική δήλωση έχει υπογραφεί και από τις δύο πλευρές και από το στρατό και από την ε, αντιπολίτευση. Όμως ε, πολλά μένουν ακόμα να γίνουν. Χρειαζόμαστε και ε, μια συνταγματική διάταξη. Μια πολύ δύσκολη και σύνθετη μετάβαση θα είναι αυτή βέβαια. Εμείς θέλουμε μια μετάβαση με μη στρατιωτική ηγεσία. Βέβαια υπάρχουν πολλές παράμετροι και ο στρατιωτικός ε, και παραστρατιωτικός κλάδος. Όλα αυτά λοιπόν αποτελούν ε, σημαντική πρόκληση, τα θέματα της λογοδοσίας, της ατιμορρησίας, σε ό,τι έχει να κάνει ιδιαίτερως και με τις επιθέσεις της 3ης Ιουνίου που ε, κόστησαν 150 ζωές στη Χαρτούμ. Είναι πολύ μεγάλες οι προσδοκίες του λαού η οικονομία βρίσκεται σε εξαιρετικά ε, δυσχερή κατάσταση μετά από χρόνια κακοδιαχείρισης ε, και απώλειας ε, εσόδων από το πετρέλαιο μετά την απόσχηση του Νοτίου Σουδάν και με μια πολύ δύσκολη κατάσταση λόγω των επιδοτήσεων. Πρέπει να υπάρξει λοιπόν ένα δίκτυο ασφαλείας. Μακροπρόθεσμα το θέμα είναι ε, η ελάφρυνση του χρέους, 60 δις ε, εθνικού χρέους που πρέπει κάπως ε, να βρεθεί μια λύση για αυτό το ζήτημα. Τι έχουμε να κάνει τώρα ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Από πολιτικής άποψης είχαμε και τον Υπουργό Εξωτερικών Πέκα Βίστο, αλλά και άλλους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η κυρία Μογκερίνη έχει συμμετάσχει ενεργά στην όλη προσπάθεια για να στηρίξει ε, την Αφρικανική Ένωση και την ε, διαμεσολάβηση της Αιθιοπίας αλλά και την συνεργασία με τις χώρες του κόλπου γιατί και αυτές δεμάτισαν κρίσιμο ρόλο. Θέλουμε λοιπόν να βρούμε μία πολιτική μετάβαση, σταθερότητα, δημοκρατία και δεύτερο βόντος για συνεργασία στον οικονομικό τομέα γιατί μπορούν να κινητοποιήσουν ε, σημαντικούς πόρους προστήριξη του Σουδάν που θα πρέπει τώρα να διοχετευτούν με έναν ανοιχτό και διαφανή τρόπο προ αυτής της δημοκρατικής μετάβασης. Οι φίλοι του Σουδάν λοιπόν ε, στη συνάντηση αυτή, αυτό είδαμε, σημειώθηκε σημαντική πρόοδος σε ό,τι αφορά τους στόχους ε, και τα μέσα προς επιτευξή τους. Το δύσκολο θα είναι η διαχείριση των προσδοκιών του λαού που επιθυμεί σταθερότητα, δημοκρατία και ευημερία. Εξαιρετικά σύνθετη βέβαια σαν διαδικασία, μακρόπνο σχέδιο, μέχρι όλα αυτά να αποφέρουν καρπούς ε, για τον πληθυσμό. Αποκινούμε συναδέλφους από την DG ε, καταρτίζουμε ένα σχέδιο στήριξης δεν θα είναι τα εκατομμύρια ή δισεκατομμύρια που μπορεί να δώσουν οι χώρες του κόλπου, αλλά σίγουρα ε, θα συμβάλλουμε σημαντικά για να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες ε, του λαού για να στηρίξουμε μια μεταβατική κυβέρνηση ε, εν ώψη και των εκλογών εντός τριετίας. Για τον Νότιο Σουδάν τώρα, όπου η εικόνα είναι λιγότερο δυναμική ή θετική. Μετά την ε, απόσχεση το 2011, αυτή η νέα χώρα ε, βρίσκεται μονίμως σχεδόν σε κατάσταση εμφυλίου πολέμου. Υπήρξε ε, μια ανανέωση της Συμφωνίας Ειρήνης, όμως τελικά δεν απέδωσε καρπούς δεν υπάρχει πραγματική πολιτική διαδικασία και εμπιστοσύνη ε, μεταξύ των πολιτικών ηγετών του Πρόεδρου Σαλβακίρ και ε, του Ρικ Μασίαρ. Υπάρχουν ε, πολιτικά παιχνίδια για να μην προχωρήσουμε προς μία ολοκληρωμένη προσέγγιση που είναι απαραίτητη για την ανοικοδόμηση της χώρας. Υποστηρίζουμε και ε, μηχανισμούς παρακολούθησης ε, της συμφωνίας και θέλουμε περαιτέρω οικονομική στήριξη, αλλά πρέπει να είμαστε πεπισμένοι πρώτα ότι ε, όλα τα μέρη θέλουν πραγματικά να συμβάλλουν σε αυτή την ενευτική διαδικασία. Υπό αυτή την αίρεση λοιπόν μπορούμε να κάνουμε περισσότερα. Ανθρωπιστική βοήθεια. Ε, φυσικά είναι πολύ σημαντικό στοιχείο ε, των ευρωπαϊκών ενεργειών ε, στην περιοχή. Θα μείνω εδώ, Πρόεδρε, και βεβαίω είμαι στη διάθεσή σα για τυχόν ερωτήσει. Ευχαριστώ κύριε Φεφάκε. Λοιπόν, να ακούσουμε ερωτήσει. Σας παρακαλώ να είστε σύντομοι συνάδελφοι. ΕΛΚ, Ευχαριστώ για την επισκόπηση που μας κάνατε, για την Αιθιοπία, το Σουδάν και το Νότιο Σουδάν και για την επίσκεψη των Μογκερίν και Νίμιτσα σε αυτή την περιοχή. Δίνουμε πολύ αναπτυξιακή βοήθεια στην Αφρική. Έχουμε τίποτα μετρήσεις για το πόσο αποτελεσματική είναι. και την αξιοποιούμε ως μέσο της διαπραγματεύσεις για την ειρήνευση. Και τι γίνεται με αυτή την ε, συμφωνία ειρήνευση στο Σουδάν. Θα κρατήσει μέχρι τις επόμενες εκλογές. Πώς το βλέπετε. Ευχαριστώ. Σοσιαλιστές. Η κυρία Αβενά. Ευχαριστώ. Για την Αιθιοπία. Είπατε ότι έχουν σημειωθεί πρόοδοι στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για τις επικείμενες εκλογές του 2020. Η πρόεδρος της ε, Εκλογικής Επιτροπής είναι πρώην ε, μέλος αντιπολίτευσης και θα ήθελα να ρωτήσω πώς βοηθάμε αυτή την Εκλογική Επιτροπή, την Κεντρική Επιτροπή Εκλογών που θα είναι βασική για να γίνουν ε, σωστά οι εκλογέ και για να υπάρξει σταθερότητα το 2020. Ευχαριστώ. Renew Europe, ο κύριος Νάρτ. Ευχαριστώ, David. Για την Αιθιοπία. Έχει ένα φιλοσοφικό σύνταγμα που επιτρέπει το δίκαιο της αυτοδιάθεσης μαζί με το Σακίτ Συνέβης. με τα νησιά είναι η μόνη χώρα που επιτρέπει αυτήν την αυτοδιάθεση αλλά η εθνότητα Συντάμα προσπαθεί να δημιουργήσει ένα δικό της κράτος στα πλαίσια της ε, Ομοσπονδίας, αλλά αυτό σημαίνει ότι το Ρώμο θα, στο Νότο θα, θα ε, διαλύει το εντελώς. Διαλύει το εντελώς. Τι μέλλον έχει η Αιθιοπία. Πώς θα μπορέσει να διατηρήσει την εσωτερική της σταθερότητα. Δεύτερον, για το Σουδάν, το Βόρειο, το, την ε, δημοκρατία του Σουδάν από την ανεξαρτησία της είναι υποστρατιωτικό καθεστώς και κυρίως από το, τη Μουχαμπαρά, τις δυνάμεις ασφαλείας. Τι μπορεί να γίνει. Ξέρετε ότι η κύρια δύναμη είναι η Σενσαγιαρουίτ και ο στρατηγός Χετμέτη που είναι εγκληματίας πολέμου. Είναι υπεύθυνο γενοκτονίας, δολοφόνος. Τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτως ώστε να μην συνεχιστεί αυτή η κατάσταση που υποτίθεται πως είναι το καθεστώς πολιτικό ενώ είναι καθεστώς των δυνάμεων ασφαλείας. Στο Νότο έχουμε φιλετικούς πολέμους μεταξύ των Νουέρ, του Σαλμπακύρ και τους Νουέρ του Μασάρ. Ξέρετε ότι ο νόμιμος πρόεδρος, πρόεδρος της χώρας, για να το πούμε έτσι, ο Σαλμπακίρ, είναι σε συμμαχία με τους Σελέκα. Με επικεφαλής τον Ουρίντ Άνταμ στην Κεντρική Αφρικανική Δημοκρατία, ο οποίος είναι ακραίο Ισλαμιστή. Τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτω ώστε ο ανύπαρκτο στην πράξη μηχανισμό ασφαλεία τη Αφρικανική Ένωση να σταματήσει να είναι αντικείμενο των δοσοληψιών και να προστατεύσει τον πληθυσμό. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο πρόεδρο. Η κυρία Φων Καμών. Για του πράσινου. Ευχαριστώ, κύριε Διευθυντά. Για τον Νότιο Σουδάν να ξεκινήσω. Το 2011 είχα την ευκαιρία μαζί με τον τότε Υπουργό Εξωτερικών Βέστερβελλε της Γερμανίας να είμαι παρούσα στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών όταν απέκτησε την ανεξαρτησία της χώρα αυτή και είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με την αντιπροσωπεία της χώρας και μας παρακάλεσε προσέξτε ακόμη και αν είναι υποδειγματική η διαδικασία απόσχησης χρειαζόμαστε πολλή στήριξη έντονη γιατί η ασφάλεια στη χώρα μας ακόμη δεν υπάρχει. Και παρακολούθησα από μακριά βέβαια την κατάσταση και η ερώτησή μου είναι μήπως ε, τη χώρα αυτή την εγκαταλείψαμε πολύ πιο γρήγορα. Μήπως τελικά τους ε, δώσαμε την ανεξαρτησία βεβιασμένα και μήπως θα μπορούσαμε να έχουμε δώσει πιο σαφή εντολή στους εκπροσώπους των ΗΠΑ για να εγγυηθούμε την ανεξαρτησία. Δεύτερη ερώτηση, η Αιθιοπία. Ναι, για πρώτη φορά μπορούμε να πούμε ότι τα πάει καλά. Αλλά, εντάξει, υπάρχουν οι βασικές ανάγκες της. Δηλαδή, ειρήνευση και επιστηστική βοήθεια. Μήπως θα πρέπει να περάσουμε στα επόμενα βήματα. Πώς θα βοηθήσουμε να υπάρξει συνεργασία, ιδιαίτερα για τις επόμενες γενιές, για να δημιουργηθούν πραγματικά προοπτικές για αυτές τις γενιές. Οικονομικές προοπτικές στο εσωτερικό της χώρας. Και ιδιαίτερα στον επιστημονικό τομέα, στην έρευνα, τι κάνετε, τι προτίθεστε να κάνετε για αυτά. Ευχαριστώ. Κύριε Φων Κραμών. Και ο κύριος Μπέργκ για τους ΙΙΝΤΕ. Ευχαριστώ. Κύριε Διευθυντά. Για τη Σομαλία θα είχα μια ερώτηση. Οι περιφερειακές εκλογές του 2019 και οι περαιτέρω εκλογές του 2020 και 2021 θεωρείτε ότι θα έχουν αρνητικό αποτέλεσμα στην Αιθιοπία και για την ευρύτερη περιοχή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Η κυρία Φωτίγκα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ για μεγάλο χρονικό διάστημα. Είχαμε πει ότι τα κοινοβουλευτικά σώματα δεν ήταν πολύ αντιπροσπευτικά. Τα λέγαμε ευγενικά αυτά. Άρα ήταν δύσκολο να δημιουργήσουμε σταθερούς δεσμούς. Αν και θεωρώ ότι η συνάντηση κορυφή του Αμπιτζάν ήταν πολύ επιτυχημένη και καρποφόρα. Πώς θα περιγράφατε το περιβάλλον που είναι αναγκαίο για να υπάρξουν παρατηρητές στις εκλογές, ιδιαίτερα στο κέρα της Αφρικής. Πρέπει οπωσδήποτε να στείλουμε παρατηρητές που να παίξουν ε, ιδιαίτερα ενεργό ρόλο. Δεύτερον, μπορείτε παρακαλώ να μας πείτε περισσότερα για τις εξελίξεις όσον αφορά την ασφάλεια σε αυτές τις χώρες. Και τι προσπάθειες κάνει η Αφρικανική Ένωση προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ πολύ ο Πρόεδρος. Και τέλος Γκουε, NGL, Βελανουέβα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Φερφάκε. Έχει νέο πρωθυπουργό εδώ και ένα χρόνο η Αιθιοπία και έτσι υπήρξε ειρήνευση με την ε, Ερυθρέα. Και υπάρχει και αυτή η δυνατότητα διαδηλώσεων και ελευθερία των μέσων. Όμως το Σαββατοκύριακο είδαμε συγκρούσεις με πάνω από 20 νεκρούς. Οπότε αυτό που μας ενδιαφέρει είναι τι θα γίνει με την εθνότητα Συντάμα που θέλει ανεξαρτησία. Θεωρείτε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να βοηθήσει να προχωρήσει αυτή η διαδικασία και να μην υπάρξουν ανησυχητικέ εξελίξεις που είδαμε το Σαββατοκυριακό. Στο Νότιο Σουδάν, μετά από ένα εμφύλιο πόλεμο πολλών ετών, υπάρχει μία ανακοχή Πρέπει να δημιουργηθεί ένα στρατός εθνικός και να σταματήσουν οι συγκρούσει για τα εσωτερικά σύνορα. Φαίνεται λοιπόν ότι δεν υπάρχουν ε, μεσολαβητές για να βοηθήσουν να σταματήσουν αυτές τις συγκρούσεις. Θα μπορούσε να παίξει πιο ενεργό ρόλο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και συγκεκριμένα, τι θα κάνουμε για τα πάνω από 2,5 εκατομμύρια προσφύγων ε, το, από τον Νότιο Σουδάν που είναι στις γύρω χώρες. Στο Σουδάν υπήρξε ένα πραξικόπημα μετά από 25 χρόνια κυβέρνησης ε, από τον Ομάρα Αλμπασίρ. Και έχουμε αυτό το μεταβατικό στρατιωτικό συμβούλιο. Δηλαδή οι ενόπλες δυνάμεις διοικούν. Είδαμε ότι υπήρξε ένα σημαντικό σημείο καμπής στις 13 Ιουλίου όταν πυροβόλησαν ε, άοπλους διαδηλωτές με πάνω από 130 νεκρούς μπροστά σε ένα στρατόνα. Υπάρχει μαζική λοιπόν καταπίεση, μας ανησυχεί. Λαμβάνουν στήριξη από τα Εμμυράτα, από την Αίγυπτο, από τη Σαουδική Αραβία, διότι τους στήριξαν. Δεν μας εκπλήττει, διότι οι σουτανικές δυνάμεις συμμετείχαν και στον πόλεμο στην Ιεμένη σε μια συνάντηση που είχαμε εδώ στις Βρυξέλλες μοιάζει να υπάρχει συμφωνία ώστε μετά από μερικούς μήνες να περάσει σε πολιτικούς η κυβέρνηση. Αλλά θα δούμε. Θα δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Και ναι, τελειώνω, τελειώνω. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπέγραψε μια συμφωνία το 2014 και έκτοτε βοηθάει την εκπαίδευση των ε, ενόπλων δυνάμεων στο Σουδάν. Έχει έννοια να κάνουν τέτοια πράγματα. Ενώ βλέπουμε ότι ο στρατός ε, καταπιέζει τον πληθυσμό. Ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστώ. Κύριε Φεφάκαρ, έχουμε άλλου δύο ομιλητέ. αν συμφωνείτε. Άλλους δύο συναδέλφους και μετά θα σταματήσουμε. Τρει. Κύριε Μίξα, Κύριε Μπένον και κύριε Πάιτ. Έκλεισε ο κατάλογο των ομιλητών. Κύριε Μίξα, ευχαριστώ μπορείτε να αναλύσετε περαιτέρω το θέμα που έχει συνέπειες σημαντικές για πολιτικές σχέσεις μεταξύ χωρών στην περιοχή, καθώς και για κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη. Τις διαφορές όσον αφορά τον επιμερισμό των υδάτων του Νείλου. Αυτό συζητήθηκε με το νέο, σε σχέση με το νέο αιθιοπικό φράγμα και τη συγκέντρωση νερού εκεί. Πώς βλέπετε τις εξελίξεις σε αυτό το τομέα. Το Ηνωμένο Βασίλειο θα έχει σήμερα νέο πρωθυπουργό. το στον Δεν θα αναφέρω τον Μπόρις, δεν θα πω τη λέξη Μπόρις. Έχουμε βάλει γραπτή ερώτηση. για τα θέματα της χρηματοδοτήσης πλευράς Ευρωπαϊκής Ενώσεως για τον έλεγχο των μεταναστευτικών ροών μέσω της διαδικασίας του Χαρτούμ. Στα ΜΜΕ είδαμε ότι έμεσα ότι θα παίρνουν κάποια, εισθετική κάποια χρήματα. Σαν ε, φορείς που παρέχουν υπηρεσίες και ενδεχομένως εμπλέκονται και στο εμπόριο μεταναστών, αυτών που έπρεπε να ελέγξουν. Έχετε σχόλιο, περιμένω την απάντηση στη γραπτή ερώτηση είχαμε τη συμφωνία για τον επιμερισμό των δυνάμεων. Αυτό είναι ένα κόλπο για να καθησυχάσουν οι διαμαρτυρίες ή είναι πραγματική η ειναι πραγματικη προσπαθεια για την Αιθιοπία. Πέρασα μερικές εβδομάδες πέρσι στην Αιθιοπία. Μίλησα σε πάρα πολλούς νέους, κυρίως ε, από φύτους μάλλον φοιτητέ, συγγνώμη, που επικρίνουν το καθεστώς. Αυτό ήταν ανεξάρτητα φιλητικής καταγωγής. Από τους ε, παλαιότερους ερχόταν οι απειλές. Ήταν ένταση μεταξύ των παλαιών και των νέων. Περισσότερο αυτό παρά μεταξύ εθνοτικών μειονοτήτων που απαρτίζουν την Αιθιοπία. Έχετε κάποιο σχόλιο πάνω σε αυτό. Ευχαριστώ. Όρμας. Πάιτ. Είναι προ συμφέρον τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω το Διεθνέ Ποινικό Δικαστήριο στο μέλλον να είναι ένα σεβαστό οργανισμός. Το Διεθνέ Ποινικό Δικαστήριο θέλει ο κύριος Αλμπασίρ να λογοδοτήσει εδώ και χρόνια. Να προσαχθεί σε αυτό το δικαστήριο. Θεωρείτε ότι στο μέλλον ε, το προβλεπόμενο θα γίνει κάτι τέτοιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να διαδραματίσει κάποιο ρόλο να ενθαρρύνει τις νέες ουδανικές αρχές ούτω ώστε να εφαρμόσουν αυτό το αίτημα, να υλοποιήσουν αυτό το αίτημα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Ευχαριστώ. Ευρύ φάσμα ερωτήσεων, κύριε Φαφάκερ. Έχετε περίπου ένα δεκάλεπτο για να απαντήσετε. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να τις ομαδοποιήσω. Είναι ο καλύτερος τρόπος αναχώρα για την Αιθιοπία. Τι συμβαίνει εκεί. Κάτι που όλο και περισσότερα συμβαίνει στην Αφρικανική Ήπειρο. Έχουμε μια νέα γενιά που ζητάει να συμμετάσχει στην οικονομική ανάπτυξη και στις θετικές διαδικασίες και τις πολιτικές εξελίξεις και να είναι κοινωνία, μια κοινωνία που εντάσσει όλους. Η Αιθιοπία είναι περιπλοκότατη χώρα λόγω της ιστορίας της και της ε, ομοσπονδιακής της δομής. Στο Σύνταγμα αναφέρεται ότι διάφορες περιοχές μπορούν να χαίρουν ενός ιδιαίτερου καθεστώτος στο ομοσπονδιακό καθεστώς. Το είδαμε στο ε, Συντάμ. Αυτό πρέπει να ε, οργανωθεί σύμφωνα με το Σύνταγμα. Αναφέρεται και δημοψήφισμα σαν ένα κομμάτι της όλης διαδικασίας. Η Αιθιοπία αντιμετωπίζει κρίσιμες στιγμές. Υπάρχει πρωθυπουργό που θέλει να κάνει σωστά πράγματα και να ξεκινήσει μεταρρυθμίσεις και έχετε όμως αντίθετες δυνάμεις. Την παλαιότερη γενιά και φυγοκεντρικές δυνάμεις, εθνοτικές, ομοσπονδιακές που έχουν περισσότερο περιθώριο και χώρο τώρα από ότι παλιά και είναι πολύ κρίσιμο θέμα, πρέπει να βρεθεί σωστή ισορροπία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αποτελεσματική και συμμετέχει στις προσπάθειες που καταβάλλονται σχετικά με αυτό. Ανέφερα τις διάφορες επισκέψεις. Έχουμε 360 εκατομμύρια ευρώ που παρέχονται φέτος και του χρόνου για υποστήριξη των μεταρρυθμίσεων που θέλει να εφαρμόσει ο Πρωθυπουργό και στον οικονομικό τομέα. Και το πρώτο που θα πρέπει να δείξει τον πληθυσμό ο Πρωθυπουργό είναι οικονομικά αποτελέσματα. Ο λαός και οι νέοι να μπορούν να έχουν μπροστά του ένα μέλλον. Προσφέρουμε υποστήριξη που σχετίζεται σαφώς με τις μεταρρυθμίσεις και το θεματολόγιο των μεταρρυθμίσεων. Αυτό που επενδύουμε λοιπόν υποστηρίζει τις παραγόμενες μεταρρυθμίσεις. Από πολιτική σκοπιά έχουμε πακέτο υποστήριξης για τις εκλογές, για την κοινωνία των πολιτών, για διάλογο μεταξύ πολιτικών κομμάτων. Συζητούμε με τη νέα επιτροπή για το, τις εκλογές και τον πρόεδρο για να το αντιμετωπίσουμε αυτό. αυτό συγγνώμη. Όταν διεξαχθούν του χρόνου οι εκλογές θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να στείλει παρατηρητές, αποστολή για παρατήρηση των εκλογών. Και έχουμε και τα αποτελέσματα των δύο προηγουμένων αποστολών που κάναμε για τις εκλογές. Έχουμε διατυπώσει κάποια σχόλια και κατευθύνσεις και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει σε τα στοιχεία για τους κινδύνους. Υφίστανται αλλά είναι και μια τεράστια ευκαιρία που παρουσιάζεται μαζί με την υποστήριξη του, στον Πρωθυπουργό θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα διάφορα θέματα με θετικό τρόπο πέραν αυτών που κάνουμε στην Αιθιοπία, αυτή κάθε αυτή. Έχουμε και περιφερειακές προσπάθειες που καταβάλλονται. Αυτό είναι κρίσιμη σημασία για την Αιθιοπία. Διασυνδεσιμότητα μεταξύ των χωρών του κέρατος Αφρικής οικονομική υποστήριξη, υποστήριξη τομέα των μεταφορών. Θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία για την περιφερειακή ασφάλεια. Όλες αυτές τις προσπάθειες κατέβαλε, είπατε εκπρόσωπος, κάθε ε, εξάμεινο συναντιόταν με τους υπουργούς και τους υπουργούς εξωτερικών των χωρών. Ε, στο Σαχέα δεν είχαμε τόσο μεγάλη επιτυχία, διότι οι χώρες χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να συντονιστούν ούτω ώστε να εμβαθυνθεί η περιφερειακή συνεργασία. Για το Σουδάν, πολλές ερωτήσεις. Τι μπορούμε να κάνουμε, τι θα συμβεί, πρέπει να διαδραματίσει σημαντικότερο, μεγαλύτερο ρόλο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Υποστηρίζουμε τη διαμεσολάβηση σε επίπεδο Αφρικής. Μόνο η Αφρικανική Ένωση κινείται σε αυτό το επίπεδο μαζί με την Αιθιοπία μέχρι τώρα έδωσαν αποτελέσματα. Ο μόνος τρόπος που μπορούμε να ενισχύσουμε το ρόλο τους είναι προσφέροντάς τους κάθε δυνατή υποστήριξη του του λεχθέντος. Παίξαμε το ρόλο μας στο Χαρτούμ, στο HIVP, μέσω του Υπουργού Εξωτερικών της Φιλανδίας. Κινηθήκαμε ερχόμενοι σε επαφή με τους θετητικούς και την αντιπολίτευση, να τους ενθαρρύνουμε να έρθουν σε επαφή και να καταλήξουν κάποια λύση. Είναι σημαντικό να ξεκινήσει η μετάβαση όσο αργή μετάβαση, η εσωτερική συνοχή τίθεται εν κινδύνο, θα προκύψουν προβλήματα, άρα ε, αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί. Παίζουμε τον ρόλο μας. Οι στατιωτικοί θα επιτρέψουν μια έναρξη μεταρρυθμίσεων. Εκεί η υποστήριξη και η συνοχή των χωρών του κόλπου είναι πάρα πολύ σημαντική στις 3 Ιουνίου όπως αναφέρθηκε ετέθη το θέμα αυτό υπάρχει κοινή αντίληψη στις χώρες του κόλπου ότι μπορούμε να έχουμε κοινό θεματολόγιο μαζί με τις χώρες του κόλπου για θέματα σταθερότητας και εκδημοκρατισμού αλλά κατανοούν οι χώρες του κόλπου ότι αν δεν υπάρχει αξιοπιστή απάντηση στις προσδοκίε του Σουδανικού λαού δεν θα υπάρξει σταθερότητα. Είναι κοινό το θεματολόγιο που οικοδομούμε και στο τέλος οι στερετικοί θα κατανοήσουν ότι υπάρχει ανάγκη για επιμερισμό τη ισχύω και να γίνει μια μετάβαση σε πολιτικό, προς πολιτικό προς διακυβέρνηση πλευράς των ε, πολιτών, των πολιτικών. Χρειάζεται χρόνος, είναι περίπλοκη η διαδικασία για να γίνει σωστή μετάβαση. Το σημαντικό είναι να ξεκινήσει η μετάβαση, να την υποστηρίξουμε και ενδεχομένως να τεθεί και η βάση για εκλογές, για την εκλογική διαδικασία. Μια διαδικασία που πρέπει να είναι αξιόπιστη. και να μπορεί να ψηφίσει ελεύθερο λαό του Σουδάν και να καταλήξει κάποια αποτελέσματα. Μόνο με κοινή προσπάθεια τα πετύχουμε όλα αυτά. Το Σουδάν, όσον αφορά τη μετανάστευση και την ασφάλεια, είναι πολύ σημαντική χώρα. Αυτοί που ρώτησαν για την υποστήριξη όσον αφορά ε, τις διάφορες, υποστήριξη διάφορες δυνάμεις και τους πολιτοφύλακες είναι ψευδείς ειδήσει αυτά που αναφέρονται επανειλημμένα τα διαψεύσαμε τα εκμεταλλεύονται διάφορες δυνάμεις οι στρατιωτικές εκεί που θέλουν να εμπλέξουν την Ευρωπαϊκή Ένωση στη διαμάχη. Δεν υπάρχει χρηματοδότηση μέχρι τώρα της Ευρωπαϊκής Ενώσης... που να έχει διοχετευτεί προς το στρατό, προς την κυβέρνηση. Δεν υπάρχουν πόροι που διοχετεύτηκαν για εκπαίδευση όσον αφορά αυτές τις, ε, τους, δυνάμει δυνάμεις στο Σουδάν. Το μόνο υποστηρίζουμε στο Χαρτούμ είναι ένα περιφερειακό κέντρο για καλύτερη διαχείριση της μετανάστευσης και στηρίζουμε τη δημιουργία δυνατοτήτων για τους δημοσίους υπαλλήλους στο Υπουργείο Εσωτερικών. Δεν υποστηρίζουμε αυτές τις δυνάμεις ταχείας υποστήριξης όπως αποκαλούνται στο Σουδάν. Για τον Νότιο Σουδάν μπορούμε να κάνουμε περισσότερα, έπρεπε να είχαμε κάνει περισσότερα. Δεν υπήρξε καλή προετοιμασία, δεν ήθελαν να οργανωμένη αυτή η απόσχηση. Οι εθνοτικές αντιθέσεις και η διαμάχη για την ισχύ στο Νότιο Σουδάν επικράτησαν. Πιέσαμε τα εμπλεκόμενα μέρη τους πιέζουμε να υπάρξει διαμεσολάβηση, προσπαθούμε να κάνουμε περισσότερα, χρειάζονται περισσότερα, κυρίως όσον αφορά τη συμφιλίωση σε τοπικό επίπεδο, αυτό εξετάζουμε περισσότερο, αναφέρθηκε από κάποιους από εσά. Χρειάζεται όμως η ηγεσία να δεσμευτεί και να επικρατήσει οικονομική διαφάνεια. Αυτό είναι απόλυτα αναγκαίο. Νομίζω ότι απάντησα στις περισσότερες ε, ερωτήσεις. Αν κάποιες λησμόνησε, με πάντα στη διάθεσή σας για να απαντήσω. Και ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Φαρφάκα. Σας ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Πολύ γόνιμη αυτή η συζήτηση. Βεβαίως αναπόκειται στους συντονιστές να αποφασίσουν πότε θα γίνει η επόμενη συνεδρίαση, αλλά θα μπορούσαμε να βάλουμε και μία επίσκεψη σε αυτή την περιοχή στο πρόγραμμά μας για το 2020-2021 και κατά την προηγούμενη θητεία είχαμε σκοπό να πάμε, τελικά δεν είναι λήφθη τέτοια απόφαση. Νομίζω όμως ότι έχει έρθει η ώρα να επισκεφθούμε την Αντίσα Ευχαριστούμε πολύ. Μας έχετε μοιράσει και ένα φυλάδιο, βλέπω. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Αφρική Φυσική σύμμαχή. Είναι στα γαλλικά βέβαια μόνο, αλλά αν σας ενδιαφέρει... Ναι, θα το στείλουμε και ηλεκτρονικά στα αγγλικά. Απλώς δεν είχαμε άλλα τυπωμένα. Όμως είναι ένα πολύ καλό φυλάδιο ε, που συντάξαμε μαζί με την ΤΕΦΚΟ συνολικά για την Αφρικανική Ήπειρο. Εξαιρετικά, σας ευχαριστούμε πολύ. Μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο θέμα της ημέρας διάταξης και θα Ladies and gentlemen, dear colleagues. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, καθίστε παρακαλώ. Για να περάσουμε στο επόμενο σημείο της μέρη της διάταξης. Συνάδελφοι, συνηθίζουμε να έχουμε καλεσμένους και να σας υποδεχόμαστε εδώ, αλλά πραγματικά θα θέλαμε να καλωσορίσουμε θερμά την κυρία Μάια Σάντου, νέα Πρωθυπουργό της Μολδαβίας, για μια ανταλλαγή απόψεων. Καλώς ήρθατε λοιπόν. Είναι μεγάλη μας χαρά που σας έχουμε εδώ και μεγάλη τιμή. Γιατί τόσοι συνάδελφοι τα τελευταία χρόνια σε αυτή την επιτροπή από τις διάφορες πολιτικές ομάδες παρακολουθούν τις εξελίξεις ε, στη χώρα σας ε, συχνά με προβληματισμό. Πολύ συχνά επίσης κάνουμε συζητήσει ε, στην ολομέλειά μας. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για τη Μολδαβία, δυστυχώς όχι πολλές φορές με θετικέ εξελίξεις, όμως τώρα είχαμε τις εκλογές στη Μολδαβία και τη νέα κυβέρνηση υπό την ηγεσία σας και τώρα σας υποδεχόμαστε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. η Επιτροπή έχει αποστείλει ε, αποστολή τριών μελών ε, στο Κίσιναου στα τέλη Ιουνίου για την υποστήριξη των ε, προσπαθειών σας. Επικεφαλής της αποστολής ήταν η κυρία Χάουταλα. Οι πολιτικές εξελίξεις είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να υλοποιηθούν Δεσμεύσει του παρελθόντο σε σχέση με τα δημοκρατικά πρότυπα, το κράτο δικαίου και την καταπολέμηση τη ε, διαφθορά, που είναι πολύ σημαντική στόχη για τη δική σα κυβέρνηση. Είναι πολύ σημαντικό να επιτευχθούν ε, αυτέ οι μεταρρυθμίσει, προκειμένου να βελτιωθούν και οι σχέσει με την Ευρωπαϊκή Ένωση και σε πολιτικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο αρρωγή Ευρωπαϊκή Ένωση και είμαι πεπισμένο ότι όλα αυτά θα καταστούν ε, δυνατά στο εγγύ μέλλον. Σας συγχαίρω και πάλι και τώρα η εξοχότητα σας έχει τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ Πρόεδρε, κύριε Μακάλιστερ, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι τιμή για μένα να είμαι η πρώτη ηγέτης τρίτη χώρας που απευθύνει το λόγο στην ε, Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων μετά τις ε, ευρωπαϊκές εκλογέ του Μαΐου. Είναι μια καλή ευκαιρία να γίνει μια ειλικρινή ανταλλαγή απόψεων για τη Μολδαβία για να συζητήσουμε τις άμεσες ε, προτεραιότητές μας και τις μακροπρόθεσμους στόχους της κυβέρνησής μας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει επικρίνει δημοσίως το προηγούμενο καθεστώς του, του οποίου ηγείται ο Ολιγάρχης Πλάκοτσουκ. Η προηγούμενη κυβέρνηση δεν σεβάστηκε σχεδόν κανένα κανόνα. Υπήρξε πλήρη πολιτικοποίηση των κυβερνητικών θεσμών, διαφθορά, ξέπλυμα χρήματο, ε, αυθαίρετε ακυρώσει εκλογών, πολιτικέ δηλώσεις, ε, πολιτικές αποφάσεις συγγνώμη, του συνταγματικού δικαστηρίου που δεν είχαν καμία λογική και δεν βασίζονταν σε γεγονότα καταδίωξη των αντιφρονούντων ε, και της ε, κοινωνίας των πολιτών, της διοίκησης των ανεξάρτητων μέσων και επιθέσεις ε, στις επιχειρήσεις. Όλα αυτά ήταν η θλιβερή πραγματικότητα στην Μολδαβία μέχρι πριν από μερικές εβδομάδες. Όλα αυτά τα κάλυπταν με φιλοευρωπαϊκή ρητορική που ελάχιστοι πίστευαν αλλά ακόμη λιγότεροι τολμούσαν να αμφισβητήσουν ανοιχτά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ποτέ δεν μάσησε τα λόγια του για τη διαφθορά του ολιγαρχικού καθεστώς στη Μολδαβία. Οι αξιολογή σας και η στήριξή σας μας βοήθησαν να επιβιώσουμε ως ε, λαός της Μολδαβίας που πιστεύει στην ελευθερία και συνεχίσαμε να αγωνιζόμαστε για την ελευθερία και σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Η διατήρηση του καθεστώτος, ε, του λιγαρικού καθεστώτος μετά τις ε, εκλογές του Φεβρουαρίου θα ήταν το χειρότερο δυνατό αποτέλεσμα γιατί θα σήμαινε ότι η Μολδοβία θα είχε καταδικαστεί να μείνει μια γκρίζα ζώνη χωρίς δημοκρατία ή ανάπτυξη με το λαό που να μην έχει καμία ελπίδα και εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση και πολλοί έφυγαν από τη χώρα. Γι' αυτό χρειάστηκε να υπάρξει ένα συνασπισμό πολιτικών δυνάμεων με αντιδιαμετρικέ απόψει πολιτικά για να μπορέσουμε να ρίξουμε αυτή την κυβέρνηση. Τα κόμματα αυτά συνεργάστηκαν επειδή η Μολδοβία ήταν σε ελεύθερη πτώση και χρειαζόταν ε, ειδική φροντίδα. Η Μολδαβία που μας την άφησε ο Πλαχονιούκ πρέπει να ξαναοικοδομηθεί από τη βάση. Σήμερα, βήμα το βήμα, διορθώνουμε και εξηγαίνουμε τη δημόσια διοίκηση και διώκονται αυτοί οι οποίοι έκλειψαν δημόσιους πόρους και εξέπλυναν χρήματα μέσω του δικαστικού και τραπεζικού συστήματος. Όλοι αυτοί θα διωχθούν. Ο βασικός στόχος της Μολδαβικής κυβέρνησης είναι η χώρα να βγει από την απόγνωση. Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα ανεξάρτητο και λειτουργικό γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα, με Γενική δηλαδή να δημιουργήσουμε κυβερνητικές ε, κυβερνητικού θεσμού που να ε, ακούνε του πολίτε να καταπολεμήσουμε τη διαφθορά, να υπάρξει δίκαιο δικαστικό σύστημα, να σταματήσει το λαθρεμπόριο και η ε, απόσυρση παράνομου εισοδήματο από τις δημόσιες ε, εταιρείες, το άνοιγμα της αγοράς σε δίκαιο ανταγωνισμό, η μεταρρύθμιση της εκπαίδευσης και της υγείας, όλα αυτά είναι οι βασικοί στόχοι της ε, τρέχουσας κυβέρνησης της χώρας. Έχουμε λοιπόν ένα ιδιαίτερα απαιτητικό καθήκον. Θέλουμε να δημιουργήσουμε μια λειτουργική δημοκρατική δημόσια διοίκηση που θα εξυπηρετεί τους πολίτες και θα ανθίσταται σε προσπάθειες να ξαναγίνει μεροληπτική. Να υπάρξει σωστός διαχωρισμός του εκτελεστικού, νομοθετικού και δικαστικού κλάδου και των οικονομικών συμφερόντων από την πολιτική. Αυτό είναι ο κοινό παρονομαστή για του πολίτε τη χώρα μα. Ανεξάρτητα από τη γλώσσα που μιλούν ή προ ποιο γεωπολιτικό μαγνητικό πόλο στρέφονται. Επανεξετάζουμε τις κυβερνητικές πολιτικές σε διάφορους τομείς. Η Μολδαβία χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται βαθιές μεταρρυθμίσεις στην δημόσια διοίκηση για να γίνει πιο αποτελεσματική, πιο επαγγελματική, πιο μεθοδική, πιο φιλική προς τους πολίτες. Ξαναξεκινήσαμε την βοήθεια από τους δωρητές και τη χρηματοδότηση που έχει παγώσει λόγω των κακών πρακτικών της προηγούμενης κυβέρνησης. Αντιμετωπίζουμε την διαφθορά και το λαθρεμπόριο στην Τρανσδρισνία που δημιουργεί απειλή για την οικονομική ασφάλεια και τη Μολδαβία και τη Ουκρανία. Επίση, έχουμε το δύσκολο καθήκον να ξανενώσουμε του πολίτε μα που έχουν ε, ε, μπει σε δύο διαφορετικέ πλευρέ ε, λόγω μια γεωπολιτική ρητορική που έβαζε του μεν κατά τον δε. Η εφαρμογή τη συμφωνία σύνδεση και τη συμφωνία ελευθέρου εμπορίου είναι η βάση τη προσπάθειά μα. Θα αξιοποιήσουμε αυτέ τι ευκαιρίε πλήρω αυτές που μας δίνονται από την πρωτοβουλία για την ε, ανατολική εταιρική σχέση ΣΥΝ για να ακολουθήσουμε την ευρωπαϊκή μας πορεία. Θέλουμε να είμαστε αξιόπιστος εταίρος και για τους πολίτες μας και για όλους τους άλλους. Δεν θα κρύψουμε τα προβλήματα, θα τα αντιμετωπίσουμε. Θέλουμε να δείτε διαφορετικά την Μολδαβία από εδώ και πέρα, ως χώρα που θέλει να γίνει όπως οι χώρες της Ένωσης, όχι στα λόγια, αλλά στην καθημερινή πρακτική της. Δεν θα παίξουμε γεωπολιτικά παιχνίδια, ούτε θα κάνουμε ανεύθυνες υποσχέσεις. Το εθνικό συμφέρον, όχι προσωπικά συμφέροντα, θα είναι η βάση της εξωτερική μας πολιτικής. Και επαναδημιουργήσαμε τη στρατηγική μας εταιρική σχέση με την Ουκρανία και τη Ρωσία. Για σχέση σχέσεις με τη Ρωσία ξαναξεκίνησε ο διάλογο που είχε ε, σταματήσει από την προηγούμενη κυβέρνηση. Αυτό δεν ήταν φυσιολογικό, γιατί έχουμε πολλά θέματα για τις διμερεί μας σχέσεις, συμπεριλαμβανομένων και θέματα διμερούς εμπορίου, που παραμένει παγωμένο. Αλλά θα είμαστε επίσης άκαμπτοι στην προστασία του εθνικού μας συμφέροντος. Θα συνεχίσουμε να πιέζουμε για να αποσυρθούν οι δυνάμεις της Ρωσίας και τα πυρομαχικά από την επικράτειά μας. Δεν θα αποδεχθούμε την ομοσπονδιοποίηση της σύγκρουσης για την Τρανσνιστρία και θα συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσει για να υπάρξει ειδικό καθεστώς για την Τρανσνιστρία εντός μιας χώρας ενιαία και κυρίαρχης, εντός των διεθνών αναγνωρισμένων συνόρων μας. Ο, ο στόχος μας είναι να μετατρέψουμε τη χώρα μας, να επανέλθει η εμπιστοσύνη των πολιτών στη χώρα και θέλουμε τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να ε, συνεχίσουμε να επιδιώκουμε να κάνουμε πραγματικότητα αυτό το όνειρο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Πρωθυπουργέ, για τα όσα μας είπατε και για το γεγονός που ότι αποδεχθήκατε την πρόσκλησή μας. Πριν δώσω το λόγο στους ε, συναδέλφους, θα ήθελα να καλωσορίσω και άλλου ε, καλεσμένου από τη Μολδαβία. Εκ δεξιών μου θα ήθελα να καλωσορίσω την νέα Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Νίκο Παπέσκου. Καλώ ήρθατε. Και βεβαίω ξέρετε τον πρέσβη, κύριο Καρά. Καλώς ήλθατε. Θα περάσουμε σε μια ανταλλαγή απόψεων. Θα ήθελα να δώσω το λόγο σε έναν εκπρόσωπο από κάθε πολιτική ομάδα, αν συμφωνείτε κι εσείς. Όμως, καλό θα ήταν να ξεκινήσουμε από την επικεφαλή τη αποστολή στη Μολδαβία πριν από δύο εβδομάδε, τη Χάιντι Χάουταλα. Από του Πρασίνου, ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, κυρία Πρωθυπουργέ. Θα ήθελα και εγώ να σας καλωσορίσω θερμά στην Επιτροπή μας. Σας ευχαριστούμε που μας αφιερώνατε χρόνο. Παρότι ήταν ε, λίγος ε, ο χρόνος, έπρεπε να τους δούμε όλους μέσα σε μια μέρα. Θέλαμε όμως το σημαντικό δυνατόν να μεταβούμε στη Μολδαβία και να ε, σας γνωρίσουμε αμέσως μετά την διαμόρφωση της κυβέρνησης. Ήδη κατέστησα σαφές ότι θα επανέλθετε στον δρόμο των μεταρρυθμίσεων και η συμφωνία σύνδεσης και η συμφωνία ελευθερών συναλλαγών ε, με ένα πιο ολοκληρωμένο πλαίσιο σίγουρα θα βοηθήσουν ε, να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας. Είπατε ότι θα επικεντρωθείτε στην μεταρρύθμιση του δικαστικού τομέα και θα ήθελα να μας ε, εξηγήσετε περαιτέρω πώς ακριβώς θα το κάνετε αυτό. Μίλησατε ξεκάθαρα και για ε, τα παραπτώματα του προηγούμενου καθεστώτος, όπως ε, το σκάνδαλο ε, διασπάθησης δημοσίου χρήματος. Δεν ήταν ε, βέβαια σαφές ε, κατά πόσο είχατε στη διάθεσή σας τα απαραίτητα έγγραφα για να εξακριβώσετε τα όσα συνέβησαν. Θα ήθελα λοιπόν να μας πείτε αν όντως τώρα έχετε συλλέξει όλα τα απαραίτητα στοιχεία και την διεθνή αυτή έκθεση και αν έχετε αναλάβει δράση. Κατά τη διάρκεια της επισκεψής μας είχε αναφερθεί ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει και έναν μηχανισμό για διακομματικό διάλογο. Διορθώστε με να κάνω λάθος, αλλά θεωρώ ότι είναι σημαντικό αυτή τη στιγμή να γεφυρώσετε ε, το χάσμα μεταξύ των ε, διαφόρων μερών προκειμένου να λειτουργήσει πιο εύρυθμα το κοινοβούλιο, μπορούμε να σας βοηθήσουμε με το λεγόμενο διάλογο Ζαμονέ προς αυτήν την κατεύθυνση. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν. Κλείνοντας θα ήθελα να χαιρετήσω την κυβέρνηση όσο έχει σχηματιστεί γιατί ε, έχει κυρίαρχη παρουσία των γυναικών και αυτό είναι κάτι το οποίο επιθυμούμε. Χρειαζόμαστε προοδευτικές γυναίκες και έτσι συμφωνούμε και με το γεγονός ότι η πλειοψηφία των μελών της κυβέρνησης είναι γυναίκες. Ευχαριστούμε Χάιντι. Πάρα πολλοί συνάδελφοι θέλουν να πάρουν το λόγο για τη Μολδαβία. Θα δώσω το λόγο σε όσους γίνεται περισσότερους. Ξεκινούμε με τον κύριο Μπαζέσκου από τη Ρουμανία. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Καλωσορίζουμε την αντιπροσωπεία από τη Μολδαβία. Θα ήθελα να τονίσω το εξής. Εδώ και 30 χρόνια η δημοκρατία της Μολδαβίας χέρι ευρωπαϊκής ε, στήριξης και εταιρικής ε, σχέσης με τη Ρουμανία. Η χώρα έχει περάσει από διάφορα στάδια, από πιο δημοκρατικές έως και λιγότερο δημοκρατικές ε, κυβερνήσεις, όπως αυτή του κ. Πλαχουτνιούκ. Όμως η χώρα ακόμα βρίσκεται σε μια γκρίζα ζώνη και η Ευρωπαϊκή Ένωση την έχει αφήσει έτσι δεν έχει δώσει μια καλή προοπτική η Ευρωπαϊκή Ένωση προς τη Μολδαβία για, ε, σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή της προοπτική. Εδώ και χρόνια ελέγχεται από, τους, ε, από δυνάμεις, από τους Ρώσους. Παρέχεται τεχνική συνδρομή για το σύστημα της δικαιοσύνης, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει παράσχει μια προοπτική ευημερία μέσω της ένταξης αυτής της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Επιτροπή μας είναι σημαντική σε ό,τι αφορά την ε, λήψη αποφάσεων πολιτικής. Γι' αυτό το των δυνατόν θα πρέπει να εξετάσουμε τη δυνατότητα η Δημοκρατία της Μολδαβίας να αποτελέσει μελλοντικά μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέσω της διαδικασίας διεύρυνσης προς Ανατολάς. Και μιλώ για αυτή την ε, διεύρυνση, γιατί ο πρόεδρος ε, Πούτιν δεν ενδιαφέρεται πια τόσο για τη Μολδαβία από ό,τι φαίνεται. Μέχρι τώρα η Τρανσδριστερία ήταν ε, μια στρατηγική σημασίας ε, ζώνη ανάσχεσης ε, για θέματα ασφαλείας ε, στην Μαύρη Θάλασσα και στην Ευρώπη. Όμως, Βλέπουμε ότι οι επιθυμίες του Προέδρου Πούτιν έχουν καλυφθεί μέσω της προσάρτησης της Κρυμαίας και εκεί έχει στρέψει την προσοχή του. Νομίζω λοιπόν ότι ο Πούτιν ε, παρουσιάζει μειωμένο, η Μολδαβία μάλλον παρουσιάζει μειωμένο ενδιαφέρον για τον Πούτιν αυτή τη στιγμή. Έχει έρθει λοιπόν η, στην κατάλληλη στιγμή να προσφέρουμε στη Μολδαβία αυτή την προοπτική της ε, προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κυρία Πύρη από τους Ελληνιστές και Δημοκράτες. I Ξέχασα πω να ανάβω το μικρόφωνο. Αυτά παθαίνει όταν λείψα το κοινοβούλιο για να κάτσει προεκλογική εκστρατεία. Ευχαριστώ. Καλώ ορίσατε, κυρία Πρωθυπουργέ. Εξ ονόματο των Σούλτσων και Δημοκρατών θα ήθελα να σα συγχαρώ και να σα ευχηθώ καλή επιτυχία με τη θητεία σας. Όπως ξέρετε, το Ευρωπαϊκό Βούλιο έχει παρακολουθήσει εκ του σύνεγγυς ε, τις εξελίξεις στη Μολδαβία κατά τη διάρκεια της τελευταίας θητείας και με μεγάλη χαρά βλέπουμε ότι έχουμε ένα νέο ξεκίνημα και εδώ στο, και στο Κισινάου. Βεβαίως, με τους ε, νέους ρόλους και αρμοδιότητες έχουμε και νέες ευθύνες και ο μολδαβικό λαός έχει ζητήσει ε, αλλαγές και μεταρρυθμίσεις που θα φέρουν την πρόοδο. Θα ήθελα να επισημάνω από την πολιτική μας ομάδα προς εσάς γιατί εμεί είμαστε γείτονες, φίλοι και σύμμαχοι. Θα σας υποστηρίξουμε αρκεί και εσείς να υλοποιήσετε το ιδιαίτερα φιλόδοξο πρόγραμμά σας και να κάνετε πραγματικότητα όλα όσα έχει ζητήσει ο λαός Μολδαβίας. Δύο ερωτήσεις. Το κόμμα των Σοσιαλιστών προσφάτως ε, κέρδισε τις εκλογές και παρότι ε, παρετήθηκε της ε, φιλοδοξίας να ηγηθεί της κυβέρνησης, ήθελαν να έχουν ε, βασικές ε, θέσεις του Υπουργικού Συμβουλίου. Ποιε ήταν οι πολιτικέ ε, προτεραιότητε τι οποίε έπρεπε να υπαναχωρήσετε για να βρεθεί κοινό έδαφο και πώ θα βρείτε την κατάλληλη ισορροπία όταν το όραμα που έχετε για τη Μολδαβία εσείς και οι σοσιαλιστές ε, είναι τελείως διαφορετικό και σε εσωτερικό και σε διεθνές επίπεδο. Ευχαριστώ. Αστραβίτσιος, εξ ονόματος ε, της ομάδας Renew Europe. Ευχαριστώ πολύ, David. Κυρία Πρωθυπουργέ, αγαπητή Μάγια, χαίρομαι πολύ που ε, σας βλέπω εδώ σε μια επίσκεψη προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με αυτή την ιδιότητα. Παλιότερα έχετε έλθει ως ε, ε, μέλος της αντιπολίτευσης αλλά τώρα βλέπουμε ότι η χώρα σας ε, έχει πλέον ε, ξεκινήσει ένα νέο κεφάλαιο. Ως ε, μόνιμος εισηγητής για τη Μολδαβία κατά την προηγούμενη θητεία, βλέπω ότι οι σχέσεις μας παραμένουν περίπλοκες με την Μολδαβία, όμως Είμαι περήφανος που το 2017 καταφέραμε να ε, βρούμε μια κοινή κατανόηση της κατάστασης ε, και να επανεξετάσουμε το θέμα της ε, μακροοικονομικής αιρεσιμότητας, παρότι είναι κάτι επώδυνο για την οικονομία σας. Είχαμε όμως βάσιμες υποψίες τότε ότι αυτά τα χρήματα δεν θα χρησιμοποιούνταν για τις ανάγκες του λαού, αλλά για τα συμφέροντα των ολιγαρχών. Συγχαρητήρια λοιπόν. Είναι βέβαια δύσκολη η θέση σας. Θεωρείται υποχείριο, κράτος υποχείριο η Μολδαβία, όπου υπάρχει ιδιαίτερα διαδεδομένη νοοτροπία διαφθοράς. και μεταξύ των πολιτικών και μια πολιτική ζωή με πολλά αρνητικά χαρακτηριστικά. Εσείς όμως ε, είστε μια σοβαρή πολιτικός που θα σταθείτε, με υπευθυνότητα όπως ε, το πράτετε και σήμερα ενώπιόν μας. Μάια, κάποια πράγματα πρέπει να γίνουν όσο γίνεται πιο σύντομα. Η μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης και του δικαστικού συστήματος. Δεν μπορούν να μείνουν τα πράγματα ως έχουν. Εμείς ε, περιμένουμε πολύ συγκεκριμένες ενέργειες ε, της μολδαβικής κυβέρνησης σε ό,τι αφορά την Ντομινίκα Μανόλια και τον ε, Μιάνο. δικαστές που κατηγορούνται για εμπλοκή σε υποθέσεις πολιτικής βαρύτητας τι είδους ε, συνδρομή θέλετε από την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να προωθήσετε τις μεταρρυθμίσεις αυτές των συντομότερο δυνατών. Σας ευχαριστώ. Παρακαλώ από τους Πρασίνους. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρωθυπουργέ. Πολύ ανοιχτή και ειλικρινή η ομιλία που κάνατε μπροστά μας. Έχω εντυπωσιαστεί πάρα πολύ. Έχω έρθει πολλές φορές στη Μολδαβία υπό την πρώτη ιδιότητά μου σαν μέλος της ε, Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΩΣΑ και, ε, και σαν μέλος της, ε, της Γερμανικού Κοινοβουλίου και της Κοινωνίας των Πολιτών μετά, ακούγοντας αυτά που έχετε να μας πείτε, ανοιχτά και ειλικρινά, πώς θέλετε γρήγορα να μεταρρυθμίσετε τη χώρα σας, με χαροποίησε. Τεράστιο όμως το έργο, Μάγια. Και περιέχονται και διάφοροι κίνδυνοι, ψηλοί κίνδυνοι θα έλεγα. Ο κίνδυνος δημιουργείται και από, το, από τον εταίρο σας στο συνασπισμό. Εξού και η πρώτη ερώτησή μας. Ποια πιθανότητα βλέπεις συνασπισμού μακράς διαρκείας κυβερνήσεως μακράς διαρκείας. Ποια είναι η εντύπωσή σου. Δεν είναι και κλεισμένον των θυρών η συνεδρίαση. Παρ' όλα αυτά όμως μπορείς να μας δώσεις μια ρελιστική απάντηση πάνω σε αυτό. Πού θα καταλήξει αυτό το εγχείρημα. Και πώς μπορεί να βοηθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και κάτι άλλο. Κάτι που ανέφερε και ο Πέτρας. Μία από τις πρώτες προτεραιότητες, κατά την άποψή μου, είναι η απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων. Μπορώ να παραθέσω διάφορα ονόματα ε, δημοσιογράφων, ακτιβιστών, αντιπολιτευομένων, δικαστών, πληροφοριοδοτών και θα ήταν σημαντικότατο το πρώτο βήμα και ένδειξη ότι το θεωρεί σοβαρό εάν αυτό αποτελέσει ύψιστη προτεραιότητα να απελευθερωθούν οι πολιτικοί κρατούμενοι. Και κάτι άλλο. τα διάφορα σκάνδαλα διαφθοράς των συνεργατών σου στο συνασπισμό. Πόσο σοβαρά θα ληφθούν υπόψη αυτά όσον αφορά το κάτω δικαίου, θέματα επιβολής του νόμου κλπ. Ποια είναι η εντύπωσή σου για όλα αυτά. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μαριάννη από το ID. Ευχαριστώ κυρία Πρωθυπουργέ. Συγχαρητήρια καταρχάς. Είχα την ευκαιρία να σας συναντήσω Συγχαρητήρια έλεγα, είχα την ευκαιρία να συναντήσω σαν εισηγητής για το σχέδιο σύνδεσης. Ήμουν εισηγητής για το Γαλλικό Κοινοβούλιο. Συγχαρητήρια για το θάρρος σας και την αντοχή σας, γιατί είναι περιπέτεια εκλογές στη χώρα σας πάντα. Άκουσα την ομιλία σας και όλοι συμφωνούμε. Υπάρχει ανάγκη κατά πολέμηση διαφθοράς που είναι μια προτεραιότητα αυτή. Μετά από αυτό όμως τι άλλο ακολουθεί. Το λέω αυτό με κάθε συμπάθεια. Σε τι συμφωνείτε όπως ρώτησε και συνάφωσα από τους Πρασίνους. Οι επαφές με τους σοσιαλιστές του κ. Νταντών. Ε, επί ποιων σημείων συμφωνείτε. Υπάρχουν και πολλά σημεία επί των οποίων διαφωνείτε και σας χωρίζουν. Ξέρετε τέλεια τους Μολδαβούς. Από ό,τι γνωρίζω περιμένουν οικονομικές μεταρρυθμίσεις οι Μολδαβοί. Ξέρετε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα σας. Η πρώτη μου ερώτηση. Επί ποιων σημείων συμφωνείτε πέρα από την καταπολέμηση της διαφθοράς που είναι πρωταρχική σημασία, και απαραίτητη. Δεύτερη ερώτηση, τι περιμένετε ακριβώς από την Ευρώπη. Διότι το πρόβλημα των θεωρήσεων ρυθμίστηκε πολύ σωστά στις μετακινήσεις στη Μολδαβία. Άκουσα ότι η Ευρώπη προτείνει πάρα πολλούς ε, πάρα πολλέ ομιλίε ε, και για το θέμα τη διαφθορά. περιμένουν επιχειρηματίε διάφορα μέτρα για τη βελτίωση του επίπεδου ζωή και την ενίσχυση των επιχειρήσεων. Σαν Πρωθυπουργό, τι έχετε να πείτε πάνω σε αυτά. Ευχαριστώ. Η κυρία Φωτίγα για το ECR. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία Πρωθυπουργέ, καλώς ήρθατε στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εγκάρδιους, εγκάρδια συγχαρητήρια για τον, ε, την ανάλυση των καθηκόντων σας. Έχω τρεις ερωτήσεις για θέματα εξωτερικών. Η κυβέρνησή σας τι στρατηγικούς και τακτικούς στόχους όσον αφορά τις διατλαντικές σχέσεις, τις σχέσεις με τις Ηνωμένε Πολιτείες και τον Καναδά, παραδείγματο χάρη, μπορείτε να βασιστείτε στην υποστήριξη του Προέδρου της χώρας πάνω σε αυτό, για θέματα ασφαλείας. Ποια είναι η κατάσταση όσον αφορά τη συνεργασία με το ΝΑΤΟ, υπάρχει γραφείο σύνδεσμο στην ε, Μολδαβία, Ποια η εξέλιξη αυτό το τομέα. Τρίτον, για ενεργειακή ασφάλεια. Ένα εύθραυστο τομέα στη Μολδαβία. Ποια είναι η κατάσταση, ποια είναι τα προβλήματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Για Γκουε, ο Χέλμουτ Σόλτ. Το λόγο ευχαριστώ Πρόεδρε. Θερμά καλωσορίζω και από την ομάδα της αριστεράς και εγώ σας χαιρετίζω Παρακολουθούσα επιμακρών τις εξελίξεις στη χώρα σας. Και πάντα θέλαμε η Μολδαβία να είναι χώρα εταίρος. Στα πλαίσια της ανατολικής γειτονίας θέλαμε να σταθερή, να προστατεύει τα συμφέροντα των πολιτών, του λαού. Συμφωνώ με πολλά από τα υποθέντα. Νομίζω ότι ο εκδημοκρατισμός της πολιτικής και κοινωνικής ζωής της χώρας σας είναι το βασικό καθήκον της νέας κυβερνήσεως. Είναι μια κυβέρνηση συνασπισμού και για μας αυτό είναι μια έκπληξη ότι ήταν εφικτός ο συνασπισμός όταν ο πρώην πρέσβης της Ευρωπαϊκής Ενώσεως είπε ότι είναι ένα χροκοπημένο κράτος η ε, Μολδαβία. Μας εκπλήσει λοιπόν το ότι επετεύχθη ο συνασπισμός. Ερώτηση. Ποιο είναι το κοινωνικό πρόγραμμα τι, που θα ακολουθήσει η κυβέρνησή σα. Πρέπει να δημιουργήσετε κλίμα εμπιστοσύνη. Εμπιστοσύνη όσον αφορά τον εκδημοκρατισμό και εμπιστοσύνη γιατί όσον αφορά την αντιμετώπιση των προβλημάτων του λαού. Να δημιουργηθεί δηλαδή η προοπτική για το μέλλον, για το λαό, να αντιμετωπιστεί η ανεργία των νέων, να αντιμετωπιστεί η φυγή εγκεφάλων που φεύγουν οι νέοι να πάνε στο εξωτερικό, η δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης σχετίζεται και με την απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων. Πρέπει να σταματήσουν οι δρομολογηθήσεις δίκες, να επικρατήσει διαφάνεια. Πώς θα υλοποιήσετε το πρόγραμμά σας, πώς θα το μεταφράσετε σε πραγματικότητα, αυτά είναι τα βασικά θέματα που μας ενδιαφέρουν για να μπορέσουμε να συνοδεύσουμε μία, ελπίζουμε, επικοδομητική και καρποφόρα πορεία που θα ακολουθήσει η κυβέρνησή σας. Σας ευχαριστώ. Αυτό ήταν ο πρώτος γύρος. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Πρωθυπουργό και μετά αν συμφωνείτε θα έχουμε δεύτερο γύρο. Πολλοί συνάδελφοι θα ήθελα να μιλήσουν. Ευχαριστώ. Ενθαρρύνθηκα από το ενδιαφέρον που δείξατε για τη χώρα μου. Σας ευχαριστώ εκ νέου, διότι μας παρατηρούσατε, μας είχατε υπόψη σας, μας δώσατε ελπίδα όταν τα πράγματα πήγαιναν πολύ άσχημα στη Μολδαβία. Δεν μιλώ μόνο για την αντιπολίτευση, για τον τρόπο που αισθανόμαστε υπό το προηγούμενο καθεστώς. Μιλάω για τους δήμαρχους, για την κοινωνία των πολιτών, για τον ανεξάρτητο τύπο. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι πέρασαν πολύ δύσκολες καταστάσεις και ήταν πραγματικά καλό και ενθαρρυντικό να γνωρίζουμε ότι τα μέλη των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων μας παρακολουθούσαν και ήξεραν τι γίνεται παρά την καλή ρητορική της προηγούμενης κυβερνήσεως. Χαίρομαι που μπορώ να απαντήσω ερωτήσεις σας μετά χαράς να ακούσω και να λάβω υπόψη συμβουλές σας. Βασική πρόκληση, όπως είπατε, είναι η μεταρρύθμιση του δικαστικού κλάδου και να δημιουργηθούν ισχυροί θεσμοί για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Δεν είμαστε αφελείς, ξέρουμε ότι αυτό δεν γίνεται μία ανοιχτή, μια τέτοια μεταρρύθμιση. Είδαμε ποια είναι η εμπειρία της Ρουμανίας Βλέπουμε πώς η Ουκρανία προς πώς προσπαθεί να δημιουργήσει θεσμούς. Προσπαθούμε να μάθουμε από την εμπειρία της Αλβανίας, από τι πρώτερε εμπειρίες της Γεωργίας. Ξέρουμε ότι δεν υπάρχει μαγική λύση. Συζητάμε πώ θα αντιμετωπίσουμε. Προχτέ, μάλιστα είχαμε μια εθνική διάσκεψη με συμμετοχή εμπειρογνωμόνων από την ε, γενικότερη περιοχή και συμμετείχαν και διάφοροι εμπλεκόμενοι τοπικοί φορείς. Θέλαμε να ενισχύσουμε την ανεξαρτησία του δικαστικού κλάδου. Από την άλλη πλευρά δεν μπορούμε να περιμένουμε ο δικαστικός κλάδος να αυτορυθμιστεί εκ των έσω, διότι δυστυχώς πολλοί από αυτούς είναι ευάλωτοι, διαφθαρμένοι, αυτοί υπηρέτησαν τα προηγούμενα καθεστώτα, διάφοροι, διάφορους πολιτικούς, άρα είναι δύσκολο πρόβλημα και αρκετοί από εσά αναφερθήκατε την απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σα. Το θέμα είναι ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να λάβει τι αποφάσει. Θα πρέπει να είναι απόφαση των δικαστών. Θα πρέπει να είναι η απόφαση των εισαγγελέων. Όπω είπα είναι αρκετά προβληματικό αυτό, διότι παρόλο που γνωρίζαμε η διαφθορά υπήρχε εκεί υπό τα προηγούμενα καθεστώτα και όχι μόνο το πρώτερο, υπό το προηγούμενο καθεστώς αυξήθηκε το πρόβλημα, αλλά εκπλήσωμε καθημερινά που ανακαλύπτω και άλλη μια διαφθορά, άλλο, άλλη μια κατάσταση διαφθοράς σε, σε κάποιο θεσμικό όργανο, σε κάποια κρατική επιχείρηση. Κατακλυζόμεθα από πληροφορίες για τη διαφθορά και η δίωξη δεν λειτουργεί ακόμα. Στέλνουμε τις πληροφορίες στην εισαγγελία. Δεν είναι ο, η που μπορεί να πάει και να συλλάβει κόσμο. Δεν μπορεί η Πρωθυπουργό, ο Υπουργό Οικονομία που ανακαλύπτει πολλά τέτοια προβλήματα διαφθοράς να ε, ξεκινήσει και να ανοίξει τέτοιες, να ανοίξει τις υποθέσεις. Είναι μεγάλο πρόβλημα και θα εκτιμούσαμε την συμβουλή σας πάνω σε αυτό, συμβουλές σας. Και περιμένουμε να βρούμε τις καλύτερες ε, λύσεις. Και πρέπει να γνωρίζετε ότι παρόλο που θέλω να λάβουν χώρα οι μεταρρυθμίσεις πολύ γρήγορα, οι προσδοκίες του λαού στη Μολδαβία είναι πάρα πολύ υψηλοί, πρέπει να το καταλάβουμε αυτό Είχαμε την απάτη στο τραπεζικό τομέα πριν από τέσσερα χρόνια, 12% του ΑΕΠ και δεν έχει ανακτηθεί ούτε μια δεκάρα από μια απάτη που αφορούσε 12% του ΑΕΠ. Και κανένας δεν έχει τιμωρηθεί για τέτοια απάτη. Ποιο θα ήθελε να ανοίξει η επιχείρηση στη Μολδαβία και πληρώσει φόρου, να ξέρει ότι οι φόροι αντί να πηγαίνουν για σχολεία, νηπιαγωγεία κλπ. πάνε για να καλύψουν τέτοιε απάτε. Άρα Υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει πολιτική βούληση, δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα. Ξέρουμε ότι είναι βασικό θέμα που έχει προτεραιότητα και θέλουμε να δούμε πώς θα κινηθούμε. Θα πρέπει να κάνουμε μια διήθηση των δικαστών και των εισαγγελέων μέσω εξωτερικού φορέα ή θα πρέπει να επιλέξουμε, επιλέξουμε άλλη προσέγγιση. Και ένα από τα βασικά προβλήματα, όπως και για το συνασπισμό, είναι ο διορισμός του νέου Γενικού Εισαγγελέα. Δεν πιστεύουμε ότι ένας άνθρωπος μπορεί να αλλάξει τα πάντα, αλλά πιστεύουμε ότι ο σωστός άνθρωπος μπορεί να ξεκινήσει την σωστή μεταρρύθμιση και ο νέος γενικός εισαγγελέα θα πρέπει να ξεκινήσει τη μεταρρύθμιση στον τομέα, να μεταρρυθμίσει την εισαγγελία, τον εισαγγελικό φορέα. Απ' την άλλη θα πρέπει να δώσει αποτελέσματα γρήγορα στις μεγαλύτερες υποθέσεις διαφθοράς που αντιμετωπίζαμε. Είναι ο μόνος ο τρόπος για να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη του λαού και να εμπιστεύεται ο κόσμο το κράτο. Συζητάμε ακόμα το θέμα. Δεν μπορώ να σα δώσω σαφέστατη απάντηση σήμερα σχετικά με το πώ θα πραγματοποιήσουμε τη μεταρρύθμιση. Αντιμετωπίζουμε το θέμα τη μη παρέμβαση, υπερβολική παρέμβαση, αυτό που μα συμβούλευε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Επί μακρόν, να μην παρεμβαίνουμε στον τομέα. Ο νόμος δίωξη που υιοθετήθηκε το 2016 επενέθηκε από όλους ετοιμάστε με γνώμονες από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους εταίρους, αλλά χρησιμοποιήθηκε το διεφθαρμένο σύστημα για να διατηρηθούν οι διεφθαρμένοι του συστήματος και να προφυλαχθούν. Εργαζόμαστε σκληρά όσον αφορά... Ε, είχαμε ετοιμάσει μια εταιρεία, μια, προσλάβουμε μια εταιρεία να ερευνήσει τον τραπεζικό τομέα και σχετικέ απάτε του τραπεζικού τομέα. Πήραμε κάποια απορίσματα κάποια παρατήματα. Δεν έχω πρόσβαση ακόμα σε όλο το κείμενο, σε όλα τα πορίσματα. Κάποιοι ισχυρίζονται ότι έχουν τα παρατήματα και έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο. Δεν μπόρεσα όμως να πείσω το Γενικό Εισαγγελέα των Τωρινό να, να κινηθεί. Και το αρμόδιο Συμβούλιο για την Ασφάλεια δεν μπόρεσε να αποφανθεί κατά πόσο οι πληροφορίες αυτές είναι ε, πραγματικές Έχω, ήρθαμε σε επαφή με την εταιρεία που έκανε την έρευνα και προσπαθούμε να ανακτήσουμε του πόρου. Ξέρετε πόσο δύσκολο να κτηθούν οι πόροι μετά από τόσα χρόνια. Θα επαναλάβω το έτοιμά μου εδώ. Οι διάφορε χώρε, οι διάφορε κυβερνήσει όπου κάποια τα χρήματα του τραπεζικού τομέα κατέληξαν, βοηθήστε από τη δική σα πλευρά να ξεκινήσουμε τι έρευνε και ελπίζουμε ότι αρκετά γρήγορα θα μπορέσουμε να έχουμε ένα γενικό εισαγγελέα που θα ξεκινήσει τις πραγματικές έρευνες από τη δική μας ε, πλευρά. Uh, Ο κύριος Μπασέσκου ανέφερε ε, τις προοπτικές ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα μας βοηθούσε πολύ κάτι τέτοιο. Καταλαβαίνουμε πρέπει να εφαρμόσουμε τη Συμφωνία Σύνδεσης. Ξέρουμε ότι επανειλημμένα οι κυβερνήσει της Μολδαβίας απογοήτευσαν τους πολίτες της χώρας αλλά και του διεθνεί εταίρου και του θεσμού τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Ξέρουμε ότι θα πρέπει να δώσουμε αποτελέσματα και να εφαρμόσουμε τρέχουσα συμφωνία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το φροντίζουμε αυτό, αλλά θα ήταν χρήσιμο να γνωρίζουμε στο τέλος ποιο θα είναι το αποτέλεσμα της σκληρής διαδικασίας που θα ακολουθηθεί θα εκτιμούσαμε την υποστήριξή σας στο διάλογο που πραγματοποιείτε. Υπήρξε μια άλλη ερώτηση σχετικά με τους συμβιβασμούς που έπρεπε να κάνουμε όταν υπογράψαμε αυτή την εταιρική σχέση. Ό,τι συμφωνήσαμε είναι δημόσιο. Η συμφωνία σύνδεσης αναφέρονται στο κυβερνητικό πρόγραμμα. Λέμε ότι η Συμφωνία Σύνδεση είναι η βάση των δραστηριοτήτων. Δεν υπάρχει κάποιο κρυμμένο θεματολόγιο. Τίποτα από αυτά που συμφωνήσαμε θα δούμε πώς θα υλοποιηθεί. Είναι δύσκολο το θεματολόγιο, δύσκολες οι μεταρρυθμίσεις. Πρέπει να κάνουμε πολλές δύσκολες μεταρρυθμίσεις. Το θεματολόγιο είναι διαφανέστατο. Είναι ένα κυβερνητικό πρόγραμμα που ψηφίστηκε υπό ιδιαίτερε ειδικέ περιστάσεις. Δεν υπήρξε καν χρόνος να συζητήσουμε την αιρεσιμότητα, τις αιρεσιμότητες, το κυβερνητικό πρόγραμμα, διότι όλα έγιναν πολύ ξαφνικά. Και νομίζω ότι ο βασικός λόγος που συνέβησαν αυτά ήταν η επιθυμία του κόσμου να απαλλαγεί από το καθεστώς, διότι το καθεστώς ήταν πολύ σκληρό και για κάποιους πολιτικούς και κάποιοι από τους πολιτικούς πιστεύω στο Συλλιστικό Κόμμα αισθάνθηκαν απειλή από το προηγούμενο καθεστώς και ήταν αποφασιστικός παράγων αυτός για να σχηματιστεί αυτού του είδους η κυβέρνηση, διότι η κυβέρνηση όπως βλέπετε είναι φιλοευρωπαϊκή οι περισσότεροι εργάστηκαν σε ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάποιοι από αυτού εργάστηκαν σε ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Είναι αφοσιωμένοι υποστηριχτέ τη Ευρώπη. Έχει αποδειχθεί χρονικά αυτό και το πρόγραμμά μας λέει σαφώς περί τίνος πρόκειται. Θέλουμε να πραγματοποιηθεί το όνειρο τη Μολδαβία η συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Σοσιαλιστικό Κόμμα έχει στενή σχέση με το Κρεμλίνο. Η κυρία Πρόεδρο ήταν εδώ πριν από μερικά λόγια. Είχαμε μια κοινή συνεδρίαση με τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου και είναι σημαντικό το Σοσιαλιστικό Κόμμα να έρθει εδώ και έτσι κι εσεί να μπορέσετε να μιλήσετε μαζί του και αυτοί να επιβεβαιώσουν εκ νέου την αποσύρωσή του στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη συμμόρφωσή του στην Συμφωνία Σύνδεση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό που ζητούν, μα ζητούν να καταβάλουμε μια προσπάθεια για βελτίωση των σχέσεων με τη Ρωσία, αλλά όπω ανέφερα στην ομιλία μου, είμαστε ανοιχτοί για να βελτιώσουμε τι οικονομικέ σχέσει με τη Ρωσία, αλλά πρέπει να σεβαστούμε και τα συμφέροντά μα και έχουμε πολλά άλλα. Θα μιλήσουμε για την ενεργειακή ασφάλεια, πρέπει να υπογράψουμε νέα σύμβαση για το φυσικό αέριο. Είναι σημαντικό για μας να καταβάλουμε προσπάθεια για να βελτιώσουμε τις ε, σχέσεις πολιτικές αιρεσιμότητες. Ήμουν εγώ που το συμβούλευα αυτό, ήταν σωστό. Αυτό μας βοήθησε να επιβιώσουμε και αυτό βοήθησε πολλούς να μην παρετηθούν από τη μάχη που έδιναν για δημοκρατία στη Μολδαβία. Διαφορετικά η επιλογή για πολλούς ανεξάρτητους δημοσιογράφους και τις κοινωνίες των πολιτών θα ήταν να φύγουν από τη χώρα. Αν αισθανόταν ότι κανείς δεν νοιάζεται για αυτά που συμβαίνουν στη Μολδαβία ή κανείς δεν κατανοεί τι συμβαίνει στη Μολδαβία. Νομίζω ότι αυτό ήταν σημαντικό και θα πρέπει να συνεχιστεί αυτό, να συνεχιστούν οι πολιτικές αιρεσιμότητες ανεξάρτητα από αυτόν που έχει την εξουσία. Αυτός είναι ένας τρόπος οι, κυβέρνηση οι κυβερνήσεις να προσέχουν και να συμπεριφέρονται σωστά. Πόσο θα κρατήσει τώρα αυτός ο κυβερνητικός συνασπισμός. Δύσκολο να σας ε, να το πω. Πραγματικά και εγώ με περιέργεια θα δω πόσο θα κρατήσει. Βεβαίω, ε, καλό θα ήταν να είναι εδώ και η πρόεδρος της Βουλής που είναι και επικεφαλής του Σοσιαλιστικού Κόμματος για να σας πει και αυτή τη γνώμη της. Αλλά <clears throat> νομίζω ότι και εκείνοι ενδιαφέρονται να κρατήσει αυτή η κυβέρνηση. Επίσης, αυτό που είναι σημαντικό είναι οι ψηφοφόροι μας, οι δικοί μας και οι ψηφοφόροι των σοσιαλιστών θέλουν να κρατήσει. Αν λοιπόν ε, τους ακούσουμε, θα κρατήσει η κυβέρνηση αρκετά για να κάνουμε μερικές οριστικές αλλαγές, για να ενισχύσουμε τις δημοκρατικές διαδικασίες και τους δημοκρατικούς θεσμούς. Αλλά έχουμε προκλήσεις, έχουμε αυτοδιοικητικές εκλογές τον ε, Οκτώβριο. Θα είναι δοκιμασία για μας να είναι ελεύθερες και τίμιες για να δείξουμε και στις, ε, στη διεθνή κοινότητα ότι μπορούμε να διοργανώσουμε τέτοιες εκλογές. Αλλά ελπίζουμε να είναι και πολιτισμένη η προεκλογική εκστρατεία. Δεν υπήρξε στο παρελθόν. Τώρα πρέπει να επιδιώξουμε να είναι πολιτισμένη. Για να μην ε, υπονομεύσει την κυβέρνηση. Βεβαίω θέλουμε να υπάρξει μια γενική εισαγγελία, ανεξάρτητη και γενικά η μεταρρύθμιση του δικαστικού κλάδου θα είναι πρόκληση. Αλλά και οι εταίροι μας λένε ότι είναι υπέρ της ανεξαρτησίας των θεσμών, της ε, εκβάθρων μεταρρύθμισης των θεσμών του κράτους. Αυτά είναι τα προβλήματα. Θα πρέπει να εργαστούμε σκληρά, να έχουμε και καλύτερη επικοινωνιακή πολιτική για να μην κάνουμε συμβιβασμούς σε τόσο σημαντικά θέματα. Γιατί αυτά είναι τα κύρια θέματα που θέσαμε. Να γίνει λειτουργικό, λειτουργικό το κράτος και, και να επανέλθει η εμπιστοσύνη των πολιτών σε αυτό. Για τα θέματα ασφάλειας, σχέση με τις Ηνωμένε Πολιτείες, τον ΝΑΤΟ, τον Καναδά. Με τις ΗΠΑ έχουμε πολύ καλή σχέση και με τον Καναδά συναντήθηκα με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ και το σχέδιο συνεργασίας με το ΝΑΤΟ λύγει, το πρόγραμμα συνεργασίας με το ΝΑΤΟ λύγει το Σεπτέμβριο και θα εκπονήσουμε νέο. Δεν υπάρχουν λοιπόν προβλήματα εκεί, παρά το ότι οι σοσιαλιστές στο παρελθόν ήταν αρνητικοί έναντι του ΝΑΤΟ. Ήταν αρνητικοί και έναντι της συμφωνίας σύνδεσης, αλλά τώρα λένε ότι είναι καλή. Αλλάζει λοιπόν ε, η επιχειρηματολογία τους και ελπίζουμε να είναι να πιστεύουν αυτά που λένε. Μας είπαν τι θα κάνουμε για τις επιχειρήσεις. Έχουμε ένα μακρύ κατάλογο ενεργειών. Συζήτησα με τις οργανώσεις των ε, εργοδοτών. Στο παρελθόν οι επιχειρήσεις υφίστανται επιθέσεις Ορισμένοι έμπαιναν φυλακή έξι μήνες, ένα χρόνο, μέχρι να δεχθούν να εκχωρήσουν τις επιχειρήσεις τους και τότε μετά τους ε, απέλυαν. Ορισμένοι λοιπόν ε, επιχειρηματίες απολύθηκαν και μας λένε τι βάσανα πέρασαν. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα της κατάργησης των μονοπωλίων, αν και μικρή χώρα έχουμε πολλά μονοπόλια. Είναι δύσκολο όμως το θέμα αυτό. Γιατί υπάρχει ένα συμβούλιο ανταγωνισμού που είναι ανεξάρτητο. Άρα δεν μπορούμε να το αλλάξουμε. Αλλά το συμβούλιο αυτό εξυπηρετεί τα μονοπόλια και βοήθησε να δημιουργηθούν. Θέλουμε λοιπόν να βελτιωθεί το επιχειρηματικό περιβάλλον, ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες. Γιατί τα άτομα αυτά έχουν ε, χαμηλό εισόδημα. Θέλουμε να δημιουργηθούν οι συνθήκες για να αυξηθούν τα εισοδήματά τους. Θέλουμε να υπάρξουν κάποια προγράμματα κατάρτισης για τους επιχειρηματίες των μικρομεσαίων, να μάθουν πώς να αναπτύξουν καλύτερα τις επιχειρήσεις τους, να κερδίσουν περισσότερα. Θέλουμε να πείσουμε και τους ε, νέους και άλλους όχι τόσο νέους ε, επιχειρηματίες στη Γαλλία, στην Ιταλία, την Ιρλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο. Θέλουμε η διασπορά να επανέλθει. Να ε, εργαστούν στη χώρα τους, κοντά στις οικογένειές τους, να δημιουργήσουν δουλειές στην Μολδαβία και καλέσαμε τη Διασπορά να επανέλθει. Μέχρι στιγμής τους προτείνουμε κρατικές θέσεις και ε, λάβαμε χίλιες αιτήσει ε, σε λιγότερο από μια εβδομάδα. Ενθαρρυντικό αυτό. Αλλά θα πρέπει να κάνουμε περισσότερα. Θα πρέπει να δείξουμε ότι υπάρχει περισσότερη ανάκαμψη για να πιστούν τα άτομα αυτά να επανέλθουν. Ενεργειακή ασφάλεια. Πολύ περίπλοκο θέμα για μας. Γιατί εξαρτώμεθα από το ρωσικό φυσικό αέριο. Ξέρετε, συζητάμε, συζητάνε μάλλον η Ρωσία και η Ουκρανία για την ε, παρεμπόδιση της ε, μεταφοράς του φυσικού αερίου μέσω της Ουκρανίας. Αν γίνει κάτι τέτοιο δεν θα μπορέσουμε να λάβουμε φυσικό αέριο από τη Ρωσία, ό,τι συμφωνία και αν έχουμε συνάψει με τη Ρωσία. Αυτό είναι πολιτικό και τεχνικό θέμα. Σήμερα αγοράζουμε φυσικό αέριο από την ε, Ρωσία σε καλύτερη τιμή από ό,τι θα μπορούσαμε να αγοράσουμε από την Ουκρανία μέσω του συστήματος αντιστροφής. Δουλεύουμε για τον αγωγό Ιασίου Κισινιό αερίου. Συνεργαζόμαστε με τις ε, ρουμανικές αρχές για να επιταχυνθεί η κατασκευή του, αλλά δεν επίκειται. Επίσης θέλουμε να διασυνδέσουμε τις ηλεκτρικές εταιρείες τις δικές μας στο, με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μέσω της Ρουμανίας. Προχωράνε αυτές οι προσπάθειες και κάποια διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα χρηματοδοτούν, αλλά θα πάρει χρόνο και αυτό, αλλά τουλάχιστον έχει ξεκινήσει. Τουλάχιστον σε μια πενταετία <clears throat> θα έχουμε εναλλακτικέ για την προμήθεια ενέργειας. Εκδημοκρατισμό. Βεβαίω, μερικά πράγματα μπορούν να γίνουν σύντομα, αλλά όχι. Για να δημιουργηθούν οι συνθήκες για την κοινωνία των πολιτών. <clears throat> για να γίνει ανεξάρτητη δημόσια δίκηση. Γιατί αυτό ήταν το κύριο όργανο των προηγουμένων κυβερνήσεων. Διότι η δημόσια δίκηση εξαρτάται εξαρτά πλήρως από το κυβερνό κόμμα. Έλεγχαν όλους τους δήμους. Θέλουμε λοιπόν η τοπική αυτοδιοίκηση και ο διοικητικός της μηχανισμός να έχει περισσότερη οικονομική αυτονομία για να είναι σημαντικό στοιχείο της δημοκρατίας και φυσικά ανεξάρτητος τύπος και κοινωνία των πολιτών. Δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει το κράτος τα ανεξάρτητα μέσα, αλλά θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να δημιουργήσουμε το κατάλληλο πλαίσιο. Για παράδειγμα, κατάργηση των μονοπωλίων για την αγορά διαφήμιση, που ήταν μεγάλο θέμα για πολλά από αυτά τα ανεξάρτητα μέσα. Και τα κοινωνικά θέματα βεβαίω, οι μικρές επιχειρήσεις. Έχουμε πολύ φτώχεια. Γι' αυτό χρειαζόμαστε οικονομική στήριξη. Για να τους στηρίξουμε. Να τους δώσουμε κάποια βοήθεια. Για, για, να, για να μπορέσουμε κατόπιν να χτίσουμε μια ισχυρή οικονομία που θα του βοηθήσει περισσότερο. Ευχαριστώ κυρία Πρωθυπουργέ. Έχετε χρόνο για ένα δεύτερο γύρο. Λοιπόν, έχει κλείσει ο κατάλογο ομιλητών για αυτό το δεύτερο γύρο. Λοιπόν, να δώσω το λόγο στου υπόλοιπου ομιλητέ. Πρώτο είναι ο κύριο Κουμπίλιο. Αλλά συγγνώμη, 1,5 λεπτό το πολύ ο καθένα. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρωθυπουργέ, αγαπητή Πρωθυπουργέ Μάια Σάντου, χαιρόμαστε που σας βλέπουμε στη θέση σας αυτή. Ξέρουμε πόσο γενναία είστε και πόσο φιλοευρωπαία αλλά ανησυχούμε για την αστάθεια του κυβερνητικού σας συνασπισμού. Αλλά είστε μεγάλη βελτίωση έναντι της προηγούμενης κυβέρνησης. Άρα θέλουμε να σας βοηθήσουμε. Εκτός από δηλώσει. πέρα από μια μακροοικονομική ενίσχυση κάποιων εκατομμυρίων, αυτό είναι το σημαντικό θέμα. Και ίσως είναι ένα ερώτημα που πρέπει να απευθύνουμε και προς τους εαυτούς μας. Διότι από την Πύρα που έχουμε από τη Λουθουανία και τη Ρουμανία που ανέφερε ο πρόεδρος Μπασέσκου, η Πύρα μας λοιπόν είναι πολύ απλή. Πρέπει να καταλάβουμε ότι οι χώρες όπως η Μολδαβία, η Γεωργία, η Ουκρανία, όπως είμαστε και εμείς παλιά, δεν μπορούμε να μεταρρυθμιστούμε από μόνοι μας επαρκώς για να προσεγγίσουμε το ευρωπαϊκό επίπεδο χωρίς μια προοπτική διεύρυνση, χωρίς ε, εμπλοκή της Ένωσης, χωρίς πραγματική εμπορική σχέση, ε, εταιρική σχέση. Άρα, τώρα που υπάρχει αυτή η νέα προσέγγιση στην ε, Ουκρανία, την Μολδαβία και τη Γεωργία, πρέπει να την αξιοποιήσουμε αυτή τη νέα ορμή. Ευχαριστώ κυρία Σάντο από τους ε, σοσιαλιστές. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κυρία Πρωθυπουργέ, Καταρχάς να σας συγχαρώ για την ανάληψη καθηκόντων σας και να σας ευχηθώ κάθε επιτυχία γιατί η επιτυχία σας θα είναι επιτυχία για όλο το λαό της Μολδαβίας. Είπατε ότι η κυβέρνησή σας θέλει η Μολδαβία να γίνει μια χώρα λογική, προβλέψιμος εταίρος, αξιόπιστος, με βάση κάποιες γεωπολιτικές αρχές. Εγώ θέλω να αναφερθώ σε δικαιώματα, ελευθερίες και εγγύησεις. Θέματα στα οποία αναφερθήκατε και εσείς είπατε ότι είναι ένα από τα κύρια μελήματα της κυβέρνησής σας. Είπατε ότι θέλετε να υπάρξει ανεξάρτητος τύπος. Αυτό είναι ανησυχία μεγάλη. <clears throat> Γιατί είναι κάτι που μας λένε πολλοί δημοσιογράφοι. Θα ήθελα να μου πείτε εάν πέρα από την κατάργηση των μονοπωλίων στην ενημέρωση και στη διαφήμιση έχετε σκεφτεί άλλα μέτρα. Επίσης Αναφερθήκατε επανειλημμένα στην κοινωνία των πολιτών, ε, τη σημασία της συμμετοχής της στην ε, δημόσια ζωή. Πρέπει, και εγώ πιστεύω, να ενισχυθεί η κοινωνία των πολιτών. Γιατί, ξέρετε, οι κοινωνίες είναι όσο δημοκρατικές, τόσο δημοκρατικές, όσο ισχυρές είναι οι κοινωνίες των πολιτών τους. Και κυρίως οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις γιατί υπάρχουν και κάποιες ε, ξένες μη κυβερνητικέ οργανώσεις που διώκονται, εξακολουθούν να διώκονται. Τι θα γίνει με αυτές τις ε, διώξεις, τις δικαστικές διώξεις. Θα μπορέσουν να συνεχίσουν να λειτουργούν ε, ικανοποιητικά. Ευχαριστώ. Ο Ούμας για το Renew. Ευχαριστώ κυρία Πρωθυπουργέ. Πολλοί παρακολουθούμε από κοντά τις εξελίξεις στη Μολδαβία. Δυστυχώς υπήρξαν πολλά σκαμπανεβάσματα. Το πιο βασικό είναι να υπάρξει κράτος δικαίου. Δεν είναι δυνατόν ε, κάθε κυβέρνηση να αλλάζει 180 μοίρες πορεία τη χώρα. Έτσι έχει γίνει τα τελευταία 10 χρόνια. Οπότε σας καλώ. Ως Πρωθυπουργός να αξιοποιήσετε τη θητεία σας για να υπάρξει μια σταθερή πορεία. Να είναι πια αυτές οι αλλαγές ανεπίστρεπτες. Ακόμη και αν η επόμενη κυβέρνηση δηλαδή έχει διαφορετικό πολιτικό προσανατολισμό να μην μπορεί να καταργήσει όλα όσα θα έχετε κάνει. Για τον ΝΑΤΟ τώρα. Προτίθεται η χώρα σας να αυξήσει το επίπεδο συνεργασίας σας με τον ΝΑΤΟ όχι μόνο έναντι τη προηγούμενη κυβέρνηση. Θέλετε να επανέλθετε στην κατάσταση πριν από 9-10 χρόνια. Και ακόμη, η Τρανσνιστρία. Τι θα κάνετε ούτως ώστε σταδιακά η επικράτεια αυτή, η περιφέρεια αυτή να έρθει πιο κοντά στην υπόλοιπη επικράτεια της ε, Δημοκρατίας της Μολδαβίας. Ευχαριστώ κύριε Σικόρσκι. Ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια, Πρωθυπουργέ. Ελπίζω να τα καταφέρετε η Μολδαβία να επανέλθει στο να είναι υπόδειγμα της ανατολικής, της ανατολικής συνεργασίας για τη σχέση με την Ένωση. Χάρηκα ιδιαίτερα που τώρα ο πρόεδρος Μπασέσκου είναι υπέρ της ένταξης της Μολδαβίας. Αν το γίνει, αν γίνει κάτι τέτοιο, θα έχουμε Ρουμάνους σε δύο έδρες στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και όχι μία που θα πρόκειται από την ενοποίηση των δύο χωρών, τη συγχώνευση. Δεύτερον, είδα πόσο διανοητικά έστασαν σαφείς για τους κινδύνους ομοσπονδιοποίησης της χώρας. Γιατί ξέρετε, θέλουν να κάνουν, ξέρετε ορισμένοι, την τρασνιστρία σαν τον Ντονμπάς. Να είναι δηλαδή ένας θύλακος που θα ελέγχεται από τους Ρώσους. Και αυτό θα αλλάξει τον γεωστρατηγικό προσανατολισμό τη χώρα. Δεν πρέπει λοιπόν να πέστε σε αυτή την παγίδα. Αλλά έχετε έλεγχο των τελωνιακών ε, αρχών για να μην είναι η τρασνιστρία δημοκρατία του λαθρεμπορίου. Και τώρα για το τραπεζικό σκάνδαλο. Ένα δις έχει βγει από το τραπεζικό σας σύστημα έχει εξαφανιστεί. Ξέρουμε πού είναι αυτά τα χρήματα και υπήρχε καμία συνενοχή ευρωπαϊκών τραπεζών και τι μπορούμε να κάνουμε για να μην επανελθεί στο μέλλον κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ. Ο κύριος Χάιζον. Σωστά το προφέρω. Χάιζον. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. ως ένας από τους λίγους συναδέλφους που μου μετέβηνε στην Μολδαβία ως ε, πολίτης, ως τουρίστας, μεταλείπεις ε, διαπίστωσα τα προβλήματα στη Μολδαβία και πόσο, πόσος χρόνος έχει σπαταληθεί ε, στην προσπάθεια να γίνεται ένα φυσιολογικό κράτος που θα μπορούσε να μπει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προ έκπληξη μου είδα τώρα ότι δημιουργήσατε αυτό το συνασπισμό με το Σοσιαλιστικό Κόμμα, όμως νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία, ίσως και μοναδική ευκαιρία με τι σημερινέ συγκυρίε, μετά από όλα τα πολιτικά διέξοδα και σκάνδαλα στη χώρα σας, να επανέλθετε σε μια σωστή πορεία για να σημειώσετε μια ευρωπαϊκή, θα έλεγα, πρόοδο. Δύο ερωτήματα. Γιατί εσείς και η κυβέρνησή σας έχετε δεσμευτεί ω προ την υλοποίηση της συμφωνία Σύνδεσης. Όμω, ε, τελικός σα στόχο είναι η ένταξή σα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δεύτερον, όπως είπαν και συνάδελφοι για τη Τρανσνιστρία. Πήγα και εκεί και είδα ότι υπάρχουν πολλές μειονότητες. Οπότε δεν είναι, πρόκειται μόνο για τους Μολδαβούς και τους Ρώσους, αλλά και άλλες ε, μειονότητες. Ποιος είναι ο τελικός ο στόχος, λοιπόν, αν έχετε κάποια επιρροή για αυτή την περιοχή. Ευχαριστώ, κυρία Τούν. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να σας εγχαρώ. Ελπίζω να κετηρίσετε το θάρρος, το κουράγιο σας ε, και την υγεία σας και όλα να πάνε καλά. Μιλήσαμε πολύ για την ε, ελευθερία του τύπου, της μη κυβερνητικέ οργανώσης. Θα ήθελα να σταθώ σε μια πολύ συγκεκριμένη υπόθεση που έχει να κάνει με τη διαφάνεια. Υπήρχε λοιπόν ένα άρθρο ε, στη Sunday Times τον Απρίλιο που ουσιαστικά στράφηκε ξεκάθαρα εναντίον μιας πολωνικής ΜΚΟ, το Open Dialogue Foundation, ε, που υπερασπίζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι κάτι το οποίο ε, κάπως στράφηκε και κατά ημού κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, χρησιμοποιήθηκε ευρέως ε, τότε κατά της ε, δημοκρατικής αντιπολίτευσης, όμως εκεί είδαμε εκ των υστέρων ότι αυτό το άρθρο βασίστηκε σε μία έκθεση που ε, εκπονήθηκε κατόπιν παραγγελίας του κυρίου Πλαχούτνιουκ παρουσιάστηκε από τα μέλη του Κοινοβουλίου που ε, ήταν πιστά σε εκείνον και σκοπός ήταν να επιτεθεί στην, ε, σε εσά και στην αντιπολίτευση που ασκούσατε τότε. Μία άλλη αποκάλυψη που έγινε μετά και ολοκληρώνω πρόεδρε ήταν ότι οι πληροφορίες που αναφέρονται σε αυτή την έκθεση προέρχονταν από την Πολωνία. Θα ήθελα λοιπόν τη βοήθειά σας. Ποιες ήταν οι πηγές. Είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον για την δημοκρατία μας. Παρακαλώ κύριε Σνάρτ. Η Μολδαβία έχει δύο σοβαρά προβλήματα. Ένα αντικειμενικό που είναι η επανίδρυση του κράτους λόγω της ε, πολιτικοποίησης του κράτους από ομάδες ε, μαφιόζικες εγκληματικές τους ολιγάρχες οπότε ελπίζω να έχετε απόλυτη συμφωνία με τους σοσιαλιστές για να προωθήσετε αυτό το στόχο. Αλλά το δεύτερο είναι οι τρομερές διαφορές σε κοινωνικό επίπεδο αλλά και στην εξωτερική πολιτική μεταξύ της, ε, του δικού σας κόμματος και του Σοσιαλιστικού Κόμματος. Βάλατε σε δεύτερη μοίρα τις διαφορές σας για να επανειδρύσετε ένα κράτος που να εξυπηρετεί τους πολίτες. <clears throat> Ειδικά για τη μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης. Μιας πραγματικής δικαιοσύνης. Και επίσης και τις άλλες εξουσίες. Έχετε την εκτελεστική και νομοθετική εξουσία, αλλά το δικαστικό σύστημα είναι απόλυτα διεφθαρμένο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τρεις συνάδελφοι από το ΕΛΚΟ, πρώτος. Μπέλτσικ. Για να Συγχαρητήρια για την εκλογή σας, ε, Πρωθυπουργέ. Αποτελείται μία νέα σελίδα στην πολιτική ζωή της Μολδαβίας και αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Εγώ σίγουρα ω μέλο τη επιτροπή για την ε, σύνδεση με την, ε, μεταξύ Μολδαβία και Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, σίγουρα εγώ θα σα στηρίξω. συμμετείχα σε πολλά προγράμματα με την προηγούμενη ιδιότητά μου ως μέλος ενός Think Tank, και θέλω να σας ρωτήσω τα εξή. Προτίθεστε να συμπεριλάβετε και την κοινωνία των πολιτών και της ΜΚΟ για την αναζωογόνηση και αναζωοπήρωση όλης αυτής της συζήτησης ε, στην εσωτερική πολιτική σκηνή. Θυμάμαι την Εθνική Σύμβαση για την Ευρωπαϊκή Ένωση στη Μολδαβία. Θα θέλατε να ξαναδιαμορφωθεί αυτό το δημόσιο βήμα που θα μπορούσε να εμπλέξει και τις ΜΚΟ στη χώρα σας. Μετά, για την ε, ε, μεταρρύθμιση του εκλογικού συστήματος που θα πρέπει να έχει γίνει εδώ και χρόνια. Ποια είναι η θέση της κυβέρνησή σας και τρίτον, αναφερθήκατε στο θέμα της ε, διασυνδεσιμότητας σε ό,τι αφορά το φυσικό αέριο. Προβλέπονται επενδύσεις σε ό,τι αφορά ε, το οδικό δίκτυο. Όχι μόνο σε σχέση με την, μάλλον σε σχέση με την Ουκρανία και, τη, και άλλες χώρε. σας χώρες. Ευχαριστώ κύριε Ραντζέλ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Αγαπητοί πρωθυπουργέ, μπορείτε να φανταστείτε τη χαρά που βιώνουμε να σας αποδεχόμαστε εδώ σήμερα ως Πρωθυπουργό μετά από όλες ε, αυτές τις συναντήσεις και στο Κισινάου και στις Βρυξέλλες. Θα έχετε διαπιστώσει λοιπόν ότι έχετε την αμέριστη υποστήριξη ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ανεξαρτήτως πολιτικής τοποθέτησης και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ένα μικρό σχόλιο μόνο, ίσως μια σύσταση. Κατανοώ πλήρως ε, το δίλημα στο οποίο βρίσκεστε για, το, για τη δικαιοσύνη, γιατί θέλετε να σεβαστείτε την ανεξαρτησία της ε, δικαιοσύνης, όμως, η δικαιοσύνη αυτή τη στιγμή δεν είναι ανεξάρτητη στη χώρα σας. Πρόκειται λοιπόν για ένα δίλημα εδώ. Να έχετε κατά νου λοιπόν ότι η κυβέρνησή σας είναι μια ματεβατική κυβέρνηση ε, μια, κατά τη διάρκεια μιας μετάβασης προς ε, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου. Και σε αυτό το πλαίσιο ίσως χρειάζεστε και την αρρωγή εξωτερικών θεσμών, Συμβούλια της Ευρώπης ή ακόμα και Ευρωπαϊκή Ένωση και θα μπορούσαμε να έχουμε ένα σχέδιο για την μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης ε, στη Μολδαβία μέσω αυτής της εξωτερικής ε, αρρωγής. Κάποιες φορές έχουμε οικονομική στήριξη, εδώ έχουμε στήριξη στο μέα του κράτους δικαίου. Αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει την κυβέρνησή σας στο έργο της. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Χαλίτσκι, τελευταίος ομιλητής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήμουν παλιότερα ε, πρόεδρος ε, της Συνόδου Πολωνίας-Μολδαβίας. Συγχαρητήρια λοιπόν και από πολωνικής πλευράς. Έχετε τη στήριξή μας. Θυμάμαι όμως ε, και το πολύ σημαντικό ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης στην μετάβαση προς τη δημοκρατία. Θυμάμαι κάποια μικρά προγράμματα αλλά πολύ αποτελεσματικά. Για την κατάσταση στην πρωτεύουσα, θεωρείτε ότι μπορεί να υπάρξουν νέε εκλογές εξαιτία ε, των εξελίξεων που είχαμε ή χρειάζεται πρώτα μία μεταρρύθμιση του ε, δικαστικού συστήματος. Ευχαριστώ πολύ. Μάια. Και πάλι πολλές ερωτήσεις. Συνάδελφοι, να ενημερώσω ότι θα υπάρξει και συζήτηση με τον Ζιλ Μπερτχόν, αλλά θα είναι πολύ σύντομη. Το αργότερο, μία παρατέταρτο, θα πρέπει να κλείσουμε τη συνεδρίαση. Έχετε λόγο για 10-15 λεπτά και μετά θα περάσουμε στο επόμενο σημείο. Ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Σε ό,τι αφορά την ισχύ και τη σταθερότητα αυτού του συνασπισμού, κατανοούμε ότι υπάρχουν ζητήματα θα ήθελα να επαναλάβω ότι δεν ήταν η χειρότερη λύση αυτού του ζητήματο. Γιατί ποια ήταν η εναλλακτική μα, να αφήσουμε το καθεστώ όπω έχει, ο κόσμο να χάσει κάθε εμπιστοσύνη ε, στη χώρα του, να φύγουν ε, οι νέοι και να μην έχουμε κανένα μέλλον για τη χώρα. Δεν υπήρχε επιλογή λοιπόν. Ξέρουμε ότι πρέπει τώρα να έχουμε γρήγορα κάποιες νίκες για να αφήσουμε τους λαϊκιστές εκτός κυβέρνησης και ταυτόχρονα να θέσουμε τις βάσεις για κάποιες μακροπρόθεσμες ε, θεσμικές μεταρρυθμίσεις. Πρέπει λοιπόν έξυπνα να συνδυάσουμε αυτά τα δύο στοιχεία και γρήγορες νίκες και μακροπρόθεσμες μεταρρυθμίσεις. Και αν έχετε συμβουλές ε, και λύσεις, είμαστε όλοι αυτιά. Για την ελευθερία του τύπου, Υπήρξε μακροσκελή συζήτηση κατά την πρώτη εβδομάδα της θητείας μου με τις ΜΚΟ αλλά και με τον τύπο. Και χαίρομαι γιατί πολλοί παρευρέθησαν. Πολλοί ε, που είχαν περάσει πολύ δύσκολα στο παρελθόν. Υπάρχει πλέον ένα σχέδιο. Θέλουμε να αλλάξουμε το οπτικοακουστικό συμβούλιο που υποτίθεται ότι είναι ανεξάρτητο, αλλά απαρτίζεται κατά κύριο λόγο από άτομα που ελέγχονται από το προηγούμενο καθεστώς. είναι ένα συμβούλιο το οποίο παίρνει τις ε, αποφάσεις ε, που επηρεάζουν ε, τον τύπο. Εμείς ζητήσαμε από τον τύπο να μας προτείνει άλλο τρόπο διορισμού των μελών της Επιτροπής που μέχρι τώρα διορίζονται από το Κοινοβούλιο, ούτως ώστε να μην επηρεάζονται από πολιτικές εξελίξεις και κόμματα. Και περιμένουμε τις προτάσεις τους προκειμένου να μην πολιτικοποιείται αυτή η διαδικασία. Το ίδιο ισχύει και για την κοινωνία των πολιτών. Πρώτα απ' όλα θέλουμε να διασφαλίσουμε τη διαφάνεια και για τον τύπο και για την κοινωνία των πολιτών. Όσο περισσότερη διαφάνεια έχουμε, τόσο διευκολύνεται και το έργο των δημοσιογράφων. Δεν χρειάζεται να περιμένουν δύο μήνε για να έχουν πρόσβαση στην πληροφορία. Δεν χρειάζεται να πληρώσουν ε, για πληροφορίε που χορηγούνται από κρατικού ε, θεσμού και δομέ. Και σίγουρα θέλουμε να εντοπίσουμε την πολιτική χρηματοδότηση ε, του τύπου με χρήματα που έχουν κλαπεί από το κράτος. Αλλά αυτό και πάλι θα το λύσει η εισαγγελία. Μιλήσατε για δίκες διεθνών ΜΚΟ. Δεν το γνωρίζω, αλλά θα το διερευνήσουμε. Ξέρουμε μόνο την περίπτωση που χρησιμοποιήθηκε εναντίον μας, ο Πλαχουτνιούκ ε, δαπάνησε πολλά χρήματα ε, για αυτή την ΜΚΟ για να μας ε, διαβάλει. Ενώ εμείς συμμετείχαμε μόνο σε μία εκδήλωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα και τα εισιτήριά μας ε, καλύφθηκαν από αυτή την ε, ΜΚΟ. Αλλά εμείς είμαστε ένα διαφανές κόμμα που χρηματοδοτείται μόνο μέσω δωρεών και αυτά ήταν χρήματα που είχαν συλλεγεί ε, νομίμως. Γι' αυτό και λαμβάνουμε χρηματοδότηση από κάποιες ΜΚΟ για να μπορούμε να συμμετέχουμε και σε ορισμένες διεθνείς τέτοιες εκδηλώσει. Για το ΝΑΤΟ θα συνεχιστεί η συνεργασία μας. Ταυτόχρονα Γνωρίζετε ότι ένα από τα μέλη του συνασπισμού μας δεν είναι υπέρμαχος του ΝΑΤΟ. Δεν θα αυξηθούν λοιπόν ιδιαίτερα οι δραστηριότητές μας, αλλά θα συνεχιστούν. Ιδίω ό,τι αφορά την επικοινωνία με το ΝΑΤΟ, γιατί στη Μολδαβία υπάρχει και πολλή προπαγάνδα που επηρεάζει την κοινή γνώμη. και η δημόσια στήριξη στην Ουκρανία, για παράδειγμα, τη ε, ε, συμμετοχή στο ΝΑΤΟ είναι πολύ χαμηλή εξαιτία τη προπαγάνδα. Γι' αυτό θέλουμε να συνεχίσουμε την εργασία, να έχουμε ένα νέο σχέδιο δράση. Δεν μπορώ να πω ότι θα αυξηθούν δραματικά ε, οι εκδηλώσεις συνεργασίας που έχουμε για τη Τρανσνιστρία να επαναλάβω και πάλι ότι το πολιτικό μας, τα πολιτικά μας κόμματα που αποτελούν το κυβερνητικό συνασπισμό είναι κατά της ε, ομοσπονδιοποίησης. Δεν ε, θεωρούμε ότι θα αποτελέσει λύση για αυτή την ε, σύγκρουση και δεν πρόκειται να την υποστηρίξουμε με κανέναν όρο και μάλιστα δεν τη χάνει και τη στήριξη των Μολδαβών. Ακόμα και αν κάποια στιγμή υπάρξει μία ε, πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο της Μολδαβίας υπέρ της ομοσπονδιοποίησης, δεν πρόκειται να προχωρήσει γιατί η πλειονότητα των Μολδαβών αντιτίθενται και κανένας πολιτικός δεν θα τολμήσει να προωθήσει μια τέτοια προσπάθεια όταν ξέρει ότι ο λαός ε, εναντιώνεται. Ποιο είναι ο σχεδιασμό μα τώρα για την Τρασνιστρία. Υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να κάνουμε, πολέμηση τη διαφθορά και του λαθρεμπορίου. Γιατί θεωρούμε ότι το οικονομικό στοιχείο τη ε, σύγκρουση είναι σημαντικό για μια πολιτική επίλυση. Αρκεί, μάλλον εφόσον κάποιοι βγάζουν εκατομμύρια εξαιτία τη διαφθορά και του λαθρεμπορίου, ε, θα είναι δύσκολο να εξευρεθεί πολιτική λύση όσο ισχύει κάτι τέτοιο. Στο παρελθόν, συνέβαινε αυτό γιατί και ε, υπήρχαν και άνθρωποι και στο Κισινάο που συμμετείχαν σε όλη αυτή τη διαπλοκή και τη διαφθορά. Τελικά είχαμε κάποιες συμφωνίες με την ε, Ουκρανία και έχουμε ήδη ζητήσει να συνεχιστεί αυτή η αποστολή UBAM στα σύνορα γιατί δεν ελέγχονται πλήρως τα σύνορα σήμερα. Υπήρξε κάποια βελτίωση τότε και μετά η Μολδαβική κυβέρνηση αποφάσισε να ανοίξει κάποια καταστήματα duty free στην Τρανιστρία και έτσι νομοποίησε το λαθρεμπόριο. Το Κοινοβούλιο την περασμένη εβδομάδα ενέκρινε ε, το νόμο με τον οποίο καταργούνται αυτά τα καταστήματα στην Τρανιστρία. Όμω, όπω είπα, το οικονομικό σκέλο είναι πολύ σημαντικό. Ε, μίλησα με τον πρόεδρο Ζελένσκι τη Ουκρανία πριν από μερικέ ημέρε και στηρίζουμε και δύο να ανοίξουν περισσότερα ε, σημεία ελέγχου συνόρων σε μια κοινή προσπάθεια με την Ουκρανία για να αντιμετωπίσουμε τη διαφθορά και το λαθρεμπόριο. Μετά έτσι θα περιοριστούν και οι πόροι του καθεστώτος και αυτό μπορεί να αλλάξει και τις ισορροπίες. Θα μπορούσε έτσι να εξευρεθεί μια πολιτική λύση. Παρότι θεωρούμε ότι αυτό θα είναι δύσκολο, δεν νομίζω ότι αυτό θα συμβεί σύντομα. γιατί όταν υπάρχει και γεωπολιτική ευκαιρία μπορεί να βρεθεί κάποια τέτοια λύση. Τέλο πάντων, εμεί θα συνεχίσουμε τι προσπάθειε όσο καλύτερα μπορούμε. Κάποιο ρώτησε κάτι άλλο. Από την απάτη, την τραπεζική που κατέξαν τα χρήματα, έχουμε έναν κατάλογο, μα τη στείλω σε όλους, όχι πολύ λεπτομερής, με τα ποσά και τις χώρες χώρες στις οποίες πήγαν τα χρήματα. Βέβαια αυτή η έκθεση και αυτός ο πίνακας χρονολογείται από παλιά, εδώ και κάποια χρόνια, μετακινήθηκαν τα χρήματα τώρα. Αυτό είναι το πρόβλημα, διότι έχει συνεχή μετακίνηση το χρήμα. Θα βρείτε τη Λετωνία όμως, Εστονία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία με μικρά ποσά, τη Ρουμανία, την Αυστρία, θα βρείτε πολλές από τις χώρες σας σε αυτόν τον κατάλογο. Πού κατέληξαν τα χρήματα. Στην Κύπρο, σε κάποιες ιδιωτικές επιχειρήσεις. Θα ήταν πολύ χρήσιμο να είχαμε κάποια βοήθεια από σας Κρίμα που πριν από δύο χρόνια, όταν αυτή η εταιρεία είχε σχέδιο για ανάκαψη των χρημάτων και το υπέβαλε στην πρώτερη κυβέρνηση, η κυβέρνηση δεν θα κάνει τίποτα, διότι τότε οι πιθανότητε ε, ανάκτηση των χρημάτων ήταν πολύ μεγαλύτερε. Το μεγαλύτερο κομμάτι του ποσού πήγε σε κάποια λετωνική τράπεζα. Αυτή η τράπεζα δεν υφίσταται πλέον και πριν από δύο χρόνια υπήρχε. Τώρα δεν ξέρουμε πού να πάμε για να ζητήσουμε τα χρήματα, διότι χρεοκόπησε η τράπεζα. Μπορούμε να σας δώσουμε τον κατάλογο και θα ήμασταν ευγνώμονες αν συνομιλούσατε με τις κυβερνήσεις σας και με τους εισαγγελείς σας και αν μας βοηθήσετε να ξεκινήσουμε τη διαδικασία από τη δική σας πλευρά για ανάκτηση. Το ίδιο για το ξέπλυμα χρήματος. Η Μολδαβία ήταν ένα τόπος όπου γινόταν ξέπλυμα χρήματος και πολλά χρήματα που ξεπλήθηκαν στη Μολδαβία μπήκαν σε λογαριασμού κάποιων τραπεζών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και καταβάλλεται σοβαρή προσπάθεια τώρα, το γνωρίζω, για να το καταπολεμήσουμε αυτό αλλά μόνοι μας δεν θα τα καταφέρουμε. Άλλη ερώτηση για την πλήρη ένταξη. Ναι, επιθυμούμε πλήρη ένταξη, αυτή είναι η ιδέα που έχουμε. Ξέρουμε ότι κάποιοι εδώ δεν θέλουν αυτό να τα ακούσουν. Γνωρίζουμε ότι πρέπει να κάνουμε πρώτα τη δουλειά μας, αλλά πιστεύω ότι αν τα καταφέρουμε, και αυτό θέλουμε, αν τα καταφέρουμε να εφαρμόσουμε όλους τους όρους, θα είμαστε σε καλύτερη θέση να έρθουμε και να ζητήσουμε τη βοήθειά σας για να προχωρήσουμε στη διαδικασία ένταξης. Εν τω μεταξύ όμως σας παρακαλώ αυτό να το θέσετε στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Αυτός είναι ο τελικός μας, ο απότερος στόχος μας. Για τη διαφάνεια και τον ανοιχτό διάλογο δεν ξέρω το πώς οι προηγούμενες αρχές έλαβαν τις πληροφορίες. Μιλήσαμε με την πρεσβεία και η πρεσβεία εκεί μας είπε ότι δεν προερχόταν οι πληροφορίες από αυτούς. Ξέρω ότι υπήρχαν κάποιες ενδείξεις που δόθηκαν, συμβουλές που δόθηκαν στην προηγούμενη κυβέρνηση να μην χρησιμοποιηθούν αυτά τα στοιχεία εναντίον μας. Συνέβη όμως, δεν έχω περισσότερες πληροφορίες, μπορώ να τις ζητήσω, γιατί είναι, ε, ίσως σας ενδιαφέρει αυτό. για τις βασικές διαφορές. Έχουμε μια συμφωνία όπου ο συνασπισμός με τους σοσιαλιστές υπεγράφει με βασικό στόχο να μην ε, υπάρχει πλέον ολιγαρχία στη χώρα, να απαλλαγούμε από τις ολιγάρχες και από τις δομές τις σχετικές. Αυτό θα χρειαστεί χρόνο. Σε κάποια φάση θα γίνουμε πολιτικοί αντίπαλοι, δεν ξέρουμε πότε, διότι είμαστε μια πολιτική δύναμη η είναι μια πολιτική δύναμη που θέλει να γίνει πιο γρήγορα η ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι σοσιαλιστές λένε δεν είναι κατά, αλλά έχουν διαφορετική, διαφορετικό χρονοδιάγραμμα που θέλουν να ακολουθήσουν. Σε κάποια φάση θα γίνουμε πολιτικοί αντίπαλοι. Είναι κανονικό αυτό, αυτό γίνεται στις χώρες όταν υπάρχουν συνασπισμοί και μετά γίνονται οι εκλογές και μετά πολεμά ένα τον άλλον για την χρήση της κοινωνίας των πολιτών και να έχουμε βήματα συζητήσεων. Κάναμε τοπικές, τομεακές μεταρρυθμίσεις όταν μια μήκυο της κοινωνίας των πολιτών ε, ζήτησε να χρησιμοποιηθεί αυτή η βάση την κοινωνία των πολιτών για τη μεταρρύθμιση του εκλογικού συστήματο. Είναι πολύ σημαντικό. Θέλουμε να αλλάξουμε το εκλογικό σύστημα. Γίνονται συζητήσει. Είμαστε γνώμονε για τη θέση σα. Τη θέση τη Επιτροπή τη Βενετία υιοθετήσαμε σε πρώτη ανάγνωση στο Κοινοβούλιο την αλλαγή του εκλογικού συστήματο. Θα γίνει ξανά αναλογικό. Λαμβάνουμε υπόψη όλε τι συστάσει τη Επιτροπή τη Βενετία και τι επόμενε ημέρε το Κοινοβούλιο θα υιοθετήσει το νέο εκλογικό νόμο στην τελική ανάγνωση Ακούσαμε την άποψη τη κοινωνία των πολιτών, θα ακούσουμε την άποψη τη διασπορά και ξέρετε ότι ήταν μεγάλο θέμα την προηγούμενη φορά. Όταν το 1 τρίτο του πληθυσμού κατοικεί στο εξωτερικό και 80% τη διασπορά ψηφίζει υπέρ τη δημοκρατία, υπέρ των φιλοδημοκρατικών κομμάτων, είναι πολύ σημαντικό αυτό να δημιουργηθούν οι συνθήκε ούτω ώστε και οι μετανάστε μα, οι ομογενεί μα να ψηφίζουν. Και σε κάποια φάση ε, θα πρέπει να επιστρέψουν αυτοί να μπορούν να επιστρέψουν βελτιώνουμε τις συνθήκες να μπορέσουν να ψηφίσουν οι ομογενείς. Για τις οδικές υποδομές υπάρχει προτεραιότητα για μας, θέλουμε να βελτιωθεί το επιχειρηματικό περιβάλλον, ανακάλυψα όμως ότι 200 εκατομμύρια ευρώ έχουν μπλοκαριστεί σε αυτή τη φάση. Χρήματα που προέρχονται από διεθνείς ε, δωρητές για την βελτίωση των ε, δρόμων λόγω κακής διακυβέρνησης κατά το παρελθόν υπήρχαν προβλήματα λόγω υποθέσεων διαφθοράς, πρέπει να πεμπλακούν αυτά τα ποσά, ούτως ώστε να λειτουργήσουν τα έργα και βέβαια θα υποβάλουμε και άλλα αιτήματα. Τώρα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αποτελεσματικά και συνετά αυτά που ήδη έχουν διατεθεί. Για τις ε, τοπικές εκλογές είχαμε πρόορες εκλογές στο Κίσινάο πέρσι και σε κάποιες άλλες ε, πόλεις διότι ο προηγούμενος ε, δήμαρχος παρετήθηκε, είχαμε πρόορες εκλογές, οι κανονικά εκλογές θα γινόταν φέτος και γι' αυτό γίνονται εκλογές φέτος. Υποτίθεται ότι θα λάμβανε χώρα τον Ιούνιο, αλλά δεν υπήρχε πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο να αποφασίσει για καθορισμό ημερομηνίας εκλογών. Τώρα οι εκλογές θα λάβουν χώρα τον Οκτώβριο και αλλάξαμε το νόμο και στο νόμο προβλέπεται πότε λαμβάνουν χώρα δημοτικέ εκλογέ ανεξάρτητα από τι πλειοψηφίε και τι αποφάσει του Κοινοβουλίου. Αυτό δεν θα είναι πλέον ε, πρόβλημα ξανά. Νομίζω ότι απάντησα σε όλε τι ερωτήσει. Πρόεδρος, νομίζω, ναι. Ήτανε πολλά αυτά που καλύψατε. Ευχαριστώ κυρία Πρωθυπουργέ που ήρθατε και μας μιλήσατε στην Επιτροπή Είμαστε Επιτροπή Εξωτικών Υποθέσεων για περίπου μια μισή ώρα. Πολλοί ομιλητέ υπογράμμισαν πόσο Χαρούμενοι ήμασταν που μπορούσαμε να σας υποδεχθούμε και ευχόμαστε και σε εσά και στην κυβέρνησή σας τον συνασπισμό ότι καλύτερο για το μέλλον της Μολδαβίας είναι πραγματικά ευρωπαϊκή χώρα η Μολδαβία και πιστεύουμε σε πολύ καλή συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ενώσεως και της μεγάλης χώρας σας, της υπέροχης χώρας σας. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρωθυπουργός. Ευχαριστώ πολύ και απευθύνω πρόσκληση σε όλους σας να επισκεφτείτε τη Μολδαβία, να μιλήσετε με τους δημοσιογράφους, με την κοινωνία των πολιτών, με τους επιχειρηματίες, με τον κόσμο στις πόλεις και στα χωριά, ούτω ώστε να δείτε μόνοι σας πόσο καλά ε, εργάζεται αυτή η κυβέρνηση και πώς τηρούμε τις υποσχέσεις που δώσαμε και σε εσά και στους πολίτες μας. Ευχαριστώ πολύ.